Mes chers collègues, euh, je vous propose de commencer notre... Ας ξεκινήσουμε τη, συνάδελφ, τη συναδρίασή μας εγκαίρως για να είμαστε ακριβείς ως συνήθως. Έχουμε καθυστερήσει κάποια λεπτά και είναι πολύ φορτωμένη η μερίσια διάταξη. Ε, tout de suite. Λοιπόν, καλό. Euh, nous allons passer au vote Ας ψηφίσουμε. Δέκα το αργότερο να ψηφίσουμε. Και ας γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία την ηλεκτρονική. Καλό λοιπόν εκείνα τα μέλη που δεν έχουν την κάρτα να φροντίσουν να τη βρουν. Και οι συνεργάτες των μελών που δεν, ε, των μελών που δεν έφτασαν να είναι σίγουροι οι βοηθοί ότι τα μέλη να μπορούν να ψηφίσουν τεχνικό πώ, να διαθέτουν την κάρτα τους με άλλα λόγια. Θα είδατε λοιπόν το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης στο κόμπι νους σας επεστάλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και διανέμεται και το κείμενο σε φυσική μορφή. Σημείο 1 λοιπόν εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη αν υπάρχουν παρατήρησεις ανακοινώσεις του Προέδρου. Είναι γραπτό στο σημείο 2, έχετε τον κατάλογο των γλωσσών. Υπάρχει μετάδοση και στο διαδίκτυο, σύθιστε. Τεράστια διεθνής ε, επιτυχία της εκπομπής αυτής. Ε, και είπα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ίγκε Γκρέσλε για τα γενέθλιά της. Inge 3 Μαρτίου δεν είναι. 2 Μαρτίου ήταν. Ξανανιώνει κάθε χρόνο ένα χρόνο λιγότερο. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά. και ο Σούριαν και Γκοντμάνης ε, ζητούν συγγνώμη που δεν μπορούν να παρίστανται και ο Νταμία Αμπάντ επίσης που έχει προσκληθεί από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας συμμετέχει σε μια σημαντικότατη εκδήλωση στη Νότια Γαλλία. Θα αφιερώσουμε μία ωρίτσα στη συζήτηση του σημείου 4, του 5 αλλά και του 6. Ήτι. Η Συντόνια θα μας παρουσιάσει στα γρήγορα ένα έγγραφο εργασίας. Πολύ σημαντικό θέμα μετά έχουμε ένα άλλο έγγραφο εργασίας θα παρουσιάσει ο Ράιμερτ η μελλοντική πρόταση σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά θα παρουσιαστεί επίσης άλλο έγγραφο εργασίας από την ΙΝΚΕ με θέμα το δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτά τα τρία σημεία είναι αλληλένδετα. Και μάλιστα τώρα που συνεχώς θα έχουμε μπροστά μας το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθέτησε και θα υποβάλει προς απόφαση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με, την, ε, με τις νέες νομικές διατάξεις και δημοσιονομικές διατάξεις ε, που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της συνθήκης της Να δώσω κατευθείαν το λόγο στη Συντόνια, αν είναι εδώ. Συντόνια, très puis Reimer, puis Inge. Και μετά στο Ράιμερ και στην Ίνγκε Και θα κάνουμε κοινή συζήτηση ξεκινώντας από την Συντόνια. Πολύ σύντομα θα κάνω μια παρουσίαση στα αγγλικά, διότι το έγγραφο συνετάχθη στα αγγλικά και δεν έχω καν την πολωνική μετάφραση. Είναι ένα συνηθισμένο βήμα στην ετήσια διαδικασία του προπολογισμού αυτό το έγγραφο που δεν είναι κάτι ασύνηθες. Σε αυτό το έγγραφο εργασίας προσπαθώ να τονίσω κάποια σημεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που παρουσιάζει τη γενική εικόνα του δημοσιονομικού προγραμματισμού βάσει της διοργανικής ε, συμφωνίας. Ως συνήθως, αυτός ο προγραμματισμός ε, δίνει ένα σχεδιασμό για το 2011, οικονομικό σχεδιασμό και αποφάσισα να ακολουθήσω το συνηθισμένο τρόπο υπογραμμίζοντας κάποιες βασικές δράσεις και κάποια βασικά κονδύλια σύμφωνα με τις διάφορες κατηγορίες του προϋπολογισμού αλλά αναφέρω και κάποιους προβληματικούς τομείς. Στόχος του εγγράφου είναι να δώσει μια συνοπτική επισκόπηση του οικονομικού προγραμματισμού, προς υπόψη σας μάλλον, αλλά απευθύνεται και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έγγραφο, γιατί περιμένω διευκρινήσεις κάποιων ζητημάτων και κάποιων σημείων που αναφέρω στα εγγραφό εργασίας θέματα που άπτονται των πιλωτικών προγραμμάτων, των προπαρασκευαστικών δράσεων και κάποιων ερωτηματικών, μεγάλων ερωτηματικών. Εντόπισα κάποια ερωτηματικά που σχετίζονται με τη στρατηγική για τη Βαλτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που κατά την άποψή μου δεν παρουσιάζεται σωστά στον όλο αυτό οικονομικό προγραμματισμό και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάποιες απαντήσεις γιατί εξακολουθεί να λείπει αυτό το στοιχείο βλέπετε σαφέστατα από αυτό τον προπολογισμό, αυτό τον οικονομικό προγραμματισμό, το πασίγνωστο πρόβλημα της οροφής. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια ελιγμών. Και αυτός ο οικονομικός προγραμματισμός ε, δείχνει αυτά τα προβλήματα. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε σε όλα τα, σώσεις κατηγορίες, σε όλα τα κεφάλαια του προπολογισμού, λεπτομερώς, δεν έχουμε χρόνο είναι αυτονόητο το έγγραφο κατά την άποψή μου. Σας παροτρύνω λοιπόν να το εξετάσετε με κριτικό μάτι και να δείτε ποια θεωρείτε σημαντικά στοιχεία. Με τα χαράς να ακούσω και διευκρινήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα σημεία που τονίζω και σε αυτή τη συνεδρίαση και στην επόμενη συνεδρίαση. Αυτά για την ώρα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Συντόνια για αυτή την παρουσίαση που ήταν πληρέστατη και πολύ σύντομη. Ο Ράιμερ τώρα. Äh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Τις τελευταίες ημέρες θα είδατε το έγγραφο εργασίας για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση με τίτλο Time to go ahead with determination, ώρα να προχωρήσουμε με επαφασιστικότητα. Βλέπω ότι είναι εδώ η Επιτροπή και ο Γενικό Διευθυντή τη, Θα ήθελα λοιπόν ίσως ε, να δω εάν μπορεί να μου απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Η Επιτροπή εχθές ενέκρινε το δημοσιονομικό πακέτο εν ώψη ε, του δημοσιονομικού πλαισίου και της διοργανικής συμφωνίας. Ε, λέγεται ότι είναι τεχνικές οι προσαρμογές. Για μένα δεν αρκούν. Δεν αρκεί να υπάρχει απλώς προσαρμογή τεχνική. Έχει όπως και να το περιγράφουμε πολιτικές επιπτώσεις και δι εν ώψη της νέας συνθήκης Λισαβόνας και των δομών της. Και βλέπω εκ πρώτης όψεως ότι έχουμε ακόμη και αλλάξει τον τίτλο της Διοργανικής Συμφωνίας για την χρηστή δημοσιονομική διοίκηση και την ε, δημοσιονομική πειθαρχία και τώρα άλλαξε ο τίτλος και λέγεται «Συνεργασία και για τα δημοσιονομικά μέτρα». Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό. Έχουμε μια διατύπωση, έναν τίτλο, τον οποίο είχαμε διαπραγματευτεί και ο οποίος δέσμευε την Επιτροπή και τον διαγράφεται επειδή υποτίθεται ότι υπάγεται στο ε, δικαίωμα της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν ισχύει, διότι είναι αντικείμενο της Διοργανικής Συμφωνίας. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε, σκοπεύουμε, πότε σκοπεύει να μας υποβάλει τις τρεις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διοργανική Συμφωνία και βέβαια πρέπει να σας επισημάνω ότι χωρίς ε, προσαρμογή, ανάλυση ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε. Αυτό λέει που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, λίγο πολύ. Και δεύτερον, για το κεφάλαιο το σχετικό με την ΚΕΠΑ, θα ήθελα να ρωτήσω πότε σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει τις προτάσεις της ε, και με βάση βέβαια τη συμφωνία για την υπηρεσία των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δημοσιονομικό δελτίο και για την τέταρτη κατηγορία και για την πέμπτη κατηγορία. Με συγκεκριμένες προτάσεις, με επαρκείς προτάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο τα ε, αριθμητικά που είχαμε στην προηγούμενη ε, περίοδο. Απλώς επαναλαμβάνω, αντιγράφτηκαν. Και Άλλη μια τελευταία ερώτηση. Σχεδόν σε όλα τα πολιετή προγράμματα έχουμε μια δέσμευση για μέσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Στα μισά της περίοδου εξετάζουμε εάν για τα τα ταμεία, για την έρευνα, για οτιδήποτε, για οτιδήποτε πολιετές πρόγραμμα, εξετάζουμε εάν πάμε καλά, αν οι στόχοι μας ε, ικανοποιούνται, πληρούνται. Έχει η Επιτροπή κάτι τέτοιο υπόψη και πότε θα γίνει αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση. Θα ήθελα πρώτα να λάβω αυτές τις απαντήσεις και μετά να συνεχίσω την παρουσίαση μου, Πρόεδρε. Καλώς σας ευχαριστώ. Σημείωσε λοιπόν η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτοιμά σας και τα ερωτήματα συντόνια. Η Ίγκε μπορεί να μας κάνει την παρουσίασή της, αν το επιθυμεί, επί του εγγράφου εργασία της. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχουμε νομίζω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία Έχουμε να κάνουμε με τα πακέτα για τις μεταβατικές διατάξεις στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Έχουμε ε, με τις δικές μου παρουσιάσεις προσπαθήσει να καταγράψουμε τι έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια, στην τελευταία μεταρρύθμιση δηλαδή, η οποία το 2007 ετέθησε ισχύ και η οποία είχε λίγο πολύ σαν στόχο να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επέτυχε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παλαιά δικά της δεινά και πάθη που προέκυψαν από τον προηγούμενο δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό το καταφέραμε λοιπόν. Από εδώ και πέρα ε, ενδέχεται να μην είναι οι δικαιούχοι, σε κάθε σημείο δηλαδή που αναφέρονται δικαιούχοι θα πρέπει να δούμε εάν και αυτοί είναι ικανοποιημένοι και αν χρειάζεται μια περαιτέρω ε, απλούστευση των ε, κανονισμών, των διατάξεων, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλή, απλή και χρηστή διαχείριση των οικονομικών μας. Υπάρχουν και κάποια στρατηγικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει σήμερα να διευκρινίσουμε, πιστεύω, και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των ε, συναδέλφων. Η αναθεώρηση που κατατέθηκε χτες, πάνω απ' όλα καταγράφει τις ε, βουλήσεις και επιθυμίες της Επιτροπής και για τις μεταφορές κονδυλίων, στα πάντα. Ε, το Συμβούλιο από την άλλη μας λέει ότι θα ήθελε μία ε, fast track, μια ταχεία διαδικασία δηλαδή για την, εξωτερική, για την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων. Μες στο μήνα μάλλον θα κατατεθεί. Δεν μας λέει η Επιτροπή λοιπόν πότε θα δούμε εμείς τις δικές μας επιθυμίες να ικανοποιούνται. Το Κοινοβούλιο πότε θα δει να ε, υποβάλλονται προτάσεις σύμφωνα με τις δικές του προτάσεις με τις δικές του επιθυμίες. Γιατί εμείς να είμαστε πάντα επεξήλου κρεμαμένοι και ποτέ να μην έχουμε την ευκαιρία να ε, εξασφαλίσουμε ικανοποίηση των ετοιμάτων μας. Ταυτόχρονα βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση για μια διαφορετική ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας των κρατών μελών για τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό πρέπει να το καθαρίσουμε σαφώς, ώστε να μην χρειάζεται στα επόμενα πέντε χρόνια να ξανάρθουμε και να το ξανασυζητήσουμε και να το, να το θεωρούμε. Επίση, θα αναφερθώ και στο άρθρο 53 του, του δημοσιονομικού κανονισμού που με πολύ σκληρό αγώνα και θα το θυμάται ο Γάιμερ πόσο πολύ είχαμε ταλαιπωρηθεί να περάσουμε τις σχετικές διατάξεις. Υπάρχουν προβλήματα και ενδέχεται να χρειαστεί να αποδεχθούμε ότι όλοι οι άλλοι παίρνουν ε, το, τη μερίδα του λέοντος, εξασφαλίζουν τα, ε, τις επιθυμητές ρυθμίσεις και για δεν έχει γίνει τίποτε. Μεγάλος κίνδυνος λοιπόν. Και αυτό το είχαμε δει και τελευταία φορά που ήταν ε, μοιρασμένε οι ψήφοι στο Συμβούλιο. Το πρόβλημα που έχουμε είναι πάντα ότι έχουμε μεγάλη πληθώρα κανόνων. Θα μπορούσαμε, και το έχω δει αυτό ήδη και το έχω επισημάνει, απλά να επιλύσουμε τα προβλήματα μειώνοντα τον αριθμό των ρυθμίσεων. Υπάρχουν πολλοί κανονισμοί, μερικέ φορέ με αντιφατικέ μεταξύ του διατάξει. Να εισαγάγουμε λοιπόν μέσα στο δημοσιονομικό κανονισμό τις ρυθμίσεις τις δημοσιονομικές των διαφόρων κανονισμών, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των διατάξεων και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας το συντονισμό ή, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγοντας την αντίφαση μεταξύ των διαφόρων διατάξεων. Τα ερωτήματα είναι πολλά λοιπόν. Ε, ξέρω βέβαια ότι αν δεν έχουμε τρόπο πίεσης, αν δεν έχουμε μέσα πίεσης, ε, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την έγκριση των δικών μας ε, τοποθετήσεων και γι' αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια να πιέσουμε. Ίσως μπορούμε, επί παραδείγματι, με την εξωτερική υπηρεσία, να τους ε, κρατήσουμε αυτούς όμοιρους. Ίσως αυτό είναι μια λύση, με κάποιο τρόπο. Ε, ναι, είμαστε πολύ διπλωμάτες όπως λέει ο Ράιμερ. Εν πάση περιπτώσει όμως αν θέλουμε κάτι να επιτύχουμε αυτή τη φορά οι δυνατότητες, τα ατού που έχουμε στα χέρια μας είναι περισσότερα από τίποτα. Επίσης, την ε, ε, χρηματοδότηση πιστώσεων για τα κτίρια. Το έχουν πει πολλοί στο παρελθόν. Ίσως αυτό είναι μια δυνατότητα. όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ήταν no-go, τα οποία το Συμβούλιο δεν δεχόταν την παραμικρή διαπραγμάτευση, μπορούμε νομίζω να τα εξασφαλίσουμε με πίεση στην υπόθεση της εξωτερικής ε, υπηρεσίας, σε παραδείγματι, για να έχουμε τις, ε, την πρόοδο που επιθυμούμε στο, στη δημοσιονομική διαχείριση. Βλέπω ότι οι συνάδελφοι ίσως κάπως μηχανία με αυτή την πρόταση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση να μην περιορίσουμε τις δικές μας επιλογές και να πιέσουμε στο βαθμό που μπορούμε για τις δικές μας θέσεις. Επίσης σημειώνω ότι έχουμε και, στον, και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχουμε την έκθεση η οποία ενδέχεται να περάσει με πολύ στενές πλειοψηφίε. Μία έκθεση πάντως, εγώ θα προτιμούσα να μην έχουμε τις δύο και έτσι καλό θα είναι να συνεργαστούμε με τον εισηγητή από εκεί ε, για να έχουμε όσο δυνατόν κοινέ συνεδριάσει όπως προτείνει, προβλέπει και ο κανονισμός για να προχωρήσουμε παράλληλα και με μία έκθεση για την απαλλαγή. Νομίζω ότι αν είμαστε προσεκτικοί και ευφυείς στην, επιλογές μας, στη συμπεριφορά μας, τα τρία αυτά ζητήματα που προανέφερα μπορούμε να τα συνδέσουμε έτσι ώστε να τα προωθήσουμε παράλληλα και τα τρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μας καλείς να προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τον αριθμό των κανόνων του δημοσιονομικού κανονισμού και στην όλη νομοθεσία και να πλουστεύσουμε και τις διαδικασίες μας. Σε μια έκθεση τίθενται τρία θέματα που στην αρχή παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο. Να επιμείνω θέλω επί της σημασίας της δουλειάς που κάνει η και του δημοσιονομικού κανονισμού. Φαίνεται ότι είναι τεχνικό ζήτημα, είναι ένα θέμα που ε, φαίνεται ότι είναι κάτι απλό, αλλά είμαστε στο επίκεντρο του κινητήρα. Παρά τις προσπάθειές της, όπως είπε, παρά τις προσπάθειες του Ράιμε, ε, που προέδρευσε της Επιτροπής Προπολογισμών, ε, είχαμε πρόβλημα από πλευρά των άλλων θεσμικών οργάνων να συμφωνήσουν με την προσέγγιση μας και έχουμε πολύ σημαντική ημερομηνία μπροστά μας ε, με τις αλλαγές που επιφέρει η συνθήκη. Λοιπόν, οι τρεις συζητητές μας εντάχει και τους ευχαριστώ για αυτό παρουσίασαν τα έγγραφα εργασίας τους που είναι έγγραφα πάρα πολύ ποιοτικά ε, μπορούμε να τα επεξεργαστούμε εποφελούμεθα από την παρουσία του κυρίου Γενικού Διευθυντού του Προπολογισμού που τον χαιρετίζω κάποια ερωτήματα του ετέθησαν ε, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει τώρα αυτή τη στιγμή σε αυτά τα ερωτήματα όμως σίγουρα έχει κάποια σχόλια να κάνει και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή ίσως για να μας συνοψίσει εν συντομία το πακέτο της Λισαβόνας που επεξεργάζεται το σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές. Πρόκειται για έγγραφα πολύ χρήσιμα και για την εργασία της Κομισιόν έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε κατά τον πλέον επικοδομητικό τρόπο στην ε, διαδικασία αυτή όπως προβλέπεται εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να απαντήσω στο αίτημά σας ε, δίδοντας και ορισμένες διευκρινήσεις θα μπορέσουμε να επανέλθουμε κατά την εξέλιξη των εργασιών. Καταρχήν θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το πακέτο που εγκρίθηκε χτες από την Κομισιόν είναι ένα πακέτο εφαρμογής της Λισαβόνας και αποκλειστικά ε, ένα τέτοιο πακέτο εφαρμογής της συνθήκης. Δηλαδή, θα παρουσιάσουμε τις προσαρμογές στον δημοσιονομικό κανονισμό που απορρέουν από την ε, εφαρμογή, από την ισχύ της συνθήκης και θα μεταμορφώσουμε τη διαθεσμική συμφωνία σε έναν κανονισμό του Συμβουλίου όπως προβλέπεται από τη συνθήκη. Τέλος, θα θέσουμε σε εφαρμογή μια νέα διαθεσμική συμφωνία για τομείς που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του Συμβουλίου και που θα πρέπει να παραμείνουν ε, στα πλαίσια της πιο ευέλικτης διαχείρισης της εργασίας μας. Δηλαδή που δεν ε, εγγράφονται, δεν ε, ενσωματώνται στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Όπως έγινε και με την προηγούμενη διαθεσμική συμφωνία. Ίσως υπάρχουν ε, καινοτόμα στοιχεία, έτσι για να το πω κάπως γραφικά, αλλά πρόκειται για μετεγγραφή ακριβώς αυτών που προαπαιτεί η συνθήκη. Και ιδιαίτερα όσον αφορά αυτόν τον ε, κανονισμό του Συμβουλίου που μεταγράφει ad hoc τα στοιχεία της ε, διαθεσμικής συμφωνίας. Πρόκειται λοιπόν για τεχνικές καθαρά προσαρμογές που γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες που απορρέουν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης. Θα επανέλθουμε σε ορισμένα ζητήματα βεβαίως που απασχολούν αυτή την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν θα σας ε, ε, διαθέσουμε την έκθεση της εκθέσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της διαθεσμικής. Δηλαδή, την αξιολόγηση της λειτουργίας του δημοσιονομικού πλαισίου που θα πρέπει να υποβάλουμε τον Απρίλιο. Κατά πάσα πιθανότητα στις 28 Απριλίου και ε, τότε θα, εγκρίνει, θα το εγκρίνει η Κομισιόν καθώς και το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011. Επίσης, σύμφωνα με τις ε, διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, θα υπάρχει μία ουσιαστική πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Και έτσι θα ανακύψει μια ανακοίνωση της Επιτροπής που θα εγκριθεί το Μάιο, κατά το δεύτερο του Μαΐου. Ε, εργάζονται εντατικά επ' αυτής οι υπεύθυνη οι της Κομισιόν. Υπάρχει και το περίφημο έγγραφο το Budget Review, για το Budget Review, για την αναθεώρηση του προπολογισμού. Δεν ήταν πλήρης η έκδοση που είχαμε μέχρι τώρα. Όπως ξέρετε, ύπτατο το Νοέμβριο, ο πρόεδρος Μπαρόζο εκφράστηκε επί του θέματος και το ίδιο και το Συμβούλιο για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτος και το φθινόπωρο θα έχουμε μία πρόταση για τους ε, ανεκτούς κινδύνους περιθώρια φάλματος. Έτσι έχει λοιπόν το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να έχετε κατά νου και εσείς και η Κομισιόν όταν εξετάζετε αυτό το έγγραφο. Και νομίζω ότι με αυτό το χρονοδιάγραμμα ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες της Επιτροπής σας καθώς και στις δικές μας ε, υποχρεώσεις όπως απορρέουν από τη συνθήκη. Ως προς τα ειδικότερα θέματα και ερωτήματα που εθίγησαν, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το θέμα του εισηγητή για το 2011 και για τη Βαλτική, η κατάσταση έχει ως εξής. Υπάρχει αυτό το εξωτερικό σκέλος με ένα εκατομμύριο ευρώ. Ε, εάν χρειαστεί θα προβλεφτούν δαπάνες με μια νομική βάση, μια νέα νομική βάση και θα πρέπει να έχουμε και σχέδια και προγράμματα. Η κατάσταση είναι απόλυτα σαφής για μένα. Από ό,τι ακούω αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν σχέδια. Υπάρχουν πολιτικές προθέσεις μόνο, όπως έχουν εκφραστεί, για κατάρτιση σχεδίων, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν υλοποιηθεί, έχει υλοποιηθεί αυτή η πολιτική θέληση με συγκεκριμένα αιτήματα προς την Κομισιόν. Από ό,τι μου λένε οι αρμόδιοι της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων και περιφερειακών υποθέσεων όταν τους ε, υπέβαλα το ερώτημα. Τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Ότι δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο. Με το χρονοδιάγραμμα λοιπόν σας έδωσα ορισμένες απαντήσεις στα ερωτήματα τουλάχιστον που έθεσε ο κύριος Μπέγκε και ίσως θα ήταν σκόπιμο να σταματήσω εδώ ε, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις των εισηγητών ή μελών της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ. Ο Ράιμερ θέλει να μιλήσει αμέσως γιατί άλλοι ζητούν το λόγο. Θέλεις να μιλήσεις τώρα, Ράιμερ. Ναι, αγαπητοί ζητώ συγγνώμη δεν είπα τίποτε ως προς το περιεχόμενο του εγγράφου εργασίας μου, εσκεμένα κατά την ε, αρχική μου τοποθέτηση, γιατί ήθελα να έχω σαφείς απαντήσεις από την Επιτροπή στα ερωτήματα αυτά. Και αν κατάλαβα καλά, η Επιτροπή τώρα σκοπεύει προς τα τέλη Απριλίου να καταθέσει μια έκθεση ως προς τον τρόπο λειτουργίας της υφιστάμενης ε, διοργανικής συμφωνίας. Ιούλιο με Σεπτέμβριο θα δούμε το έγγραφο για την, δημοσιονομ... για την αναθεώρηση του κανονισμού, Bachelor review. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής δεν είπε τίποτα για το τι σκοπεύει να κάνει ως προς το δημοσιονομικό δελτίο του σχετικό με τη Λισαβόνα, τις εξελίξεις, τι θα συμπεριλάβει μέσα, στην, ε, μέσα στον κανονισμό στις προτάσεις για το 2011, για τις πολυετείς προοπτικές ή θα το πάει μετά το 2013. Και επίση δεν είπε τίποτα για το τι σκοπεύει να κάνει ως προς την κοινή ευθύνη που έχουμε αναλάβει για την, μακρο... για την μέσο πρόθεσμη αναθεώρηση. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά και πάλι να επανέλθω πρόεδρε για να κάνω τις προτάσεις μου. Ε, Ωραία. Γέρα, θέλεις να παρέμβεις τώρα, διότι ο Ράιμερ θα προτιμούσε να παρέμβει πρώτα ο Γενικός Διευθυντής, εκτός και αν έχεις μία συμπληρωματική. Γέραν, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Γι' αυτό ήθελα να παρέμβω τώρα. Κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα σαφές είναι ποιες είναι οι προθέσεις της Κομισιόν σε σχέση με τους αρχικούς στόχους της ε, ε, αναθεώρησης, της ενδιάμεσης αναθεώρησης, διότι μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο προϋπολογισμό 2011, 2012 και 2013, δεν υπάρχουν περιθώρια. Εδώ έχουμε έξι διαφορετικά πακέτα μία πρόταση για τον προϋπολογισμό 2011 για το δημοσιονομικό κανονισμό για τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013. Τι θα γίνει όμως σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση τη στιγμή που θα αναθεωρήσουμε και τις οροφές 2011-2013. Θα το δούμε ως όλον, ως συνολική πρόταση 2011-2013 για τις υπόλοιπες δημιουσυνοτικές προοπτικές ή θα το δούμε ξεχωριστά στις ακροάσεις των Επιτρόπων. Από πλευράς Επιτροπής μας ζητήσαμε μία πρόταση για την ενδιάμεση αναθεώρηση πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και θα ήθελα να μου το διασαφηνίσει ακόμα περισσότερο η Κομισιόν τι προθέσεις έχει. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για μας και για την φετινή διαδικασία του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ, Γκέραν. Υπάρχουν και δύο άλλοι συντονίστες που ζήτησαν το λόγο για να συμπληρωθούν οι ερωτήσεις προς την Κονσιόν. Ο Σαλβαδόρ και μετά η, η Χέλγκα. Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ. Απλώς να συμπληρώσω αυτά που προελέχθησαν, νομίζω ότι η Κομισιόν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τις ακροάσεις των επιτρόπων. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ορισμένε ενδείξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επερχόμενες προτάσεις για την ενδιάμεση αναθεώρηση διότι θα επηρεάσουν όχι μόνο τη διαδικασία προετοιμασίας του προϋπολισμού 2011, αλλά και τις επικείμενες συζητήσεις στις πολιτικές ομάδες για να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση για την χρηματοδότηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Θεωρώ λοιπόν αυτή την ε, καθυστέρηση απαράδεκτη. Θα ήθελα η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την υποβολή προτάσεων για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Υπάρχει και το εκρεμές ζήτημα για το πότε η Επιτροπή θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της για να μας υποβάλει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για τις εξωτερικές δράσεις. Διότι θέλει να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που είναι ένα θέμα κλειδί για μας για να μπορέσουμε να δεχτούμε τα μέτρα και τις προτάσεις εξωτερικών δράσεων και με το, την πρόταση δημοσιονομικού κανονισμού θα ξέρουμε ποιες θα είναι και οι προθεσμίες για το προσχέδιο προϋπολογισμού. Από όσο γνωρίζω, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί με το πρώτο στο πρώτο ορόσημο, δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου. Είμαστε ήδη στο Μάρτιο, γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε πότε θα μας υποβάλλετε αυτό το προσχέδιο. Ευχαριστούμε Σαλβαδόρ. Μας εκπλήσει αυτό το ε, αίτημα όπως εκφράστηκε. Η Χέλγα, τι έχει να μας πει εκείνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο ίδιο θέμα θα τοποθετηθώ και εγώ όπως και ο προλαλής σας για να υπενθυμίσω ότι είχαμε και τη Συμφωνία για τις μεσονομικές προοπτικες Προοπτικές 2007-2013 ναι. με σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση που μάλιστα σήμαινε αναλυτικά αναφερόταν και στα, στα έσοδα και στις δαπάνες. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε τότε σε επίπεδο Συμβουλίου λάβει δεσμεύσεις από τον τότε Υπουργό Προεδρεύοντα ε, της Αυστρίας. Τη δέσμευση λοιπόν φαντάζομαι ότι είναι και ακόμη το Συμβούλιο. Η Επιτροπή όμως, η Επιτροπή θα έπρεπε να διεκδικεί τη θέση της στο, ε, στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα έπρεπε να είναι εκείνη που θα έσπροχνε προς τέτοιου είδους ε, αναθεωρήσεις για να μπορεί να διατηρήσει και το δικαίωμα της πρωτοβουλίας της θα έπρεπε να καταθέτει τέτοιες προτάσεις. Κανονικά θα έπρεπε να το έχει πράξει το 2009. Τώρα έχουμε φτάσει στο Μάρτιο του 2010, διάφορα non-papers λοιπά μπορεί να έχουμε δει, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις με σαφείς έννοιες, με αντίληψη αυτή της κατάστασης δεν έχουμε δει. Και γι' αυτό παρακαλώ να είμαστε όλοι οι συνάδελφοι σαφείς προς την Επιτροπή και να μην ε, αφήνουμε με ρητορίες να περνάει αναπάντητα τα ερωτήματά μας. Συγκεκριμένες δεσμεύσεις θέλουμε. Τι θα κάνει, μέχρι πότε, σε ποιο βαθμό και εάν θα υπάρχουν εξελίξει από το 2013 και μετά ή αν θα παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο. Γιατί εδώ θα ήθελα να επισημάνω και τα όσα είπε ο Μπαρόσο ότι δε, και σε σχέση με αυτά να πω ότι η στάση της Επιτροπής δεν στέκει πολιτικά δεν έχει συνάφεια με τις δεσμεύσεις του Μπαρόσο. Εάν θέλουμε μια νέα πολιτική, εάν θέλουμε μια Ευρώπη για τον πολίτη, εάν θέλουμε μια ουσιαστική πολιτική πρέπει να έχουμε σαφείς δεσμεύσεις και για τον προπολογισμό πάνω απ' όλα. Και από αυτό περιμένω να ακούσω κάτι από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Έλγα. Ο Γενικός Άκουσα τις παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων που είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι. Διότι βλέπουν ότι πια δεν υπάρχουν περιθώρια ως προς τις οροφές. Έχετε περιθώρια έκφρασης εσείς για την, ε, ως προς την κατάρτιση των ε, προτάσεων της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η Κομισιόν, όπως είπα και πριν, θα υποβάλει μία έκθεση για τη λειτουργία της διαθεσμικής συμφωνίας και με προτάσεις, με τις ε, κατάλληλες προτάσεις. Αν τώρα με ρωτάτε τώρα τι περιθώρια έχουμε, για την υποβολή προτάσεων δεν μπορώ να σας πω τίποτα, διότι είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί από το Διευθυντήριο των Επιτρόπων. Γίνονται εργασίες σε επίπεδο υπηρεσιών, η δημοσιονομική κατάσταση είναι γνωστή. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι εργασίας για να ανταποκριθούμε σε τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα. Θα το αποφασίσει το Διευθυντήριο Επιτρόπων, εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ. Υπογραμμίζω όμως ότι θα έχετε αυτή την έκθεση με τις ε, προτάσεις στις 28 Απριλίου, μαζί με την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2011. σε σχέση με την αναθεώρηση του προγράμματος, όπως ε, είπε και ο κύριος Μπέγκε, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αναλάβει δεσμεύσεις επί του θέματος και πέραν από τις γενικές διατάξεις, διατάξεις γενικής αξιολόγησης που υπάρχουν στο δημοσιονομικό κανονισμό, όπου η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα μέσα. Ε, έχουμε τη διαχείριση του, του συστήματος με βάση τις δράσεις, activity-based management. Προβλέπουμε και θέλουμε να δούμε τι απαιτήσει υπάρχουν ως προς την αξιολόγηση. Πρόκειται όμως για προγράμματα τα οποία ε, ενέκρινε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δηλαδή για αυτές τις αξιολογήσεις. Εγκρίθηκαν λοιπόν αυτά τα προγράμματα αξιολόγηση σύμφωνα με τις ε, διατάξεις και εμείς θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών. Όσον αφορά τις εξωτερικές υπηρεσίες, θα λάβετε Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας ε, πω πιο συγκεκριμένα, αλλά το ταχύτερο δυνατόν θα λάβετε ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, όπου θα λαμβάνονται υπόψη, θα λαμβάνονται υπόψη η εφαρμογή αυτής, ε, η, μάλλον η αρχή της δράσης αυτής της υπηρεσίας εξωτερικών σχέσεων. Συνεργαζόμαστε με την κυρία Άστον για το θέμα αυτό. Έχει επιτελεστεί πρόοδος. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν μετά από συζήτηση των ε, γενικών μας πολιτικών την 11η Μαρτίου θα εγκρίνουμε τις προτάσεις τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού και τις τροποποίησεις των κανόνων σε σχέση με τον κανονισμό. Μετά την 11η Μαρτίου όλα αυτά. Άρα τις μετέπειτα εβδομάδες θα λάβετε τις προτάσεις μας. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία ως προς την έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε και εμείς να προχωρήσουμε γρήγορα. Και η κυρία Άστον ε, έχει πρωταρχικό μέλημα να προχωρήσει αρκετά γρήγορα, έτσι ώστε να έχουμε υποδομές για τις εξωτερικές αυτές υπηρεσίες, για να μπορέσουν να αναλάβουν δράση το ταχύτερο δυνατόν. Ενοποιημένα δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα υποβάλει ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού κατά τις επόμενες εβδομάδες. Αυτά μπορώ να σας πω ως προς το θέμα αυτό. Ως προς το ερώτημα της κυρίας, της κυρίας ε, για την ενδιάμεση αναθεώρηση και για το, μιλάμε για την διαθεσμική συμφωνία ε, για αυτήν ήδη σας είπα, ξέρετε την ημερομηνία, το Διευθυντήριο θα αποφασίσει για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, με βάση τις διαπιστώσεις που θα γίνουν ως προς την ε, κατάσταση του προϋπολογισμού, ως προς την δημοσιονομική αναθεώρηση, την ενδιάμεση αναθεώρηση, αν λάβουμε υπόψη την ιδιάζουσα κατάσταση, της Επιτροπής που διαχειρίστηκε το όλο θέμα πέρσι τον Νοέμβριο. Αναβάλαμε την ημερομηνία έγκρισης, τη μεταθέσαμε μάλλον και ο πρόεδρος Επιτροπής θεωρεί ότι η ημερομηνία στόχος και αυτό νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ημερομηνία λοιπόν στόχος για την παρουσίαση αυτού του εγγράφου θα έπρεπε να είναι ο Ιούλιος του τρέχοντος έτους. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Γι' αυτό και ακριβώς είπα στην προηγούμενη μου παρέμβαση ότι ίσως γίνει κάτι τέτοιο ή τον, ή τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Νομίζω λοιπόν ότι απάντησα στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην αυτή σειρά παρεμβάσεων. Ε, Ευχαριστούμε, Γενική. Ε, Ράιμερ. Ο Ράιμερ. Δείχνει βέβαια όλη η συζήτηση ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο έχουμε δει τους τελευταίους μήνες ως στάση. Ότι ιδιαίτερα η πτυχή της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης στη διοργανική συμφωνία, συμφωνία, στις δημοσιονομικές προοπτικές, ερμηνεύεται διαφορετικά από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, από ότι όχι μόνο εμείς θεωρούμε, αλλά από ότι βλέπουμε να έχει γίνει η διαπραγμάτευση στο παρελθόν. Αλλάζει δηλαδή ε, ερμηνεία. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είναι, είναι τα ζητήματα, τα θέματα δύσκολα και περίπλοκα όντω. αλλά ταυτόχρονα στην αναθεώρηση, στην αναθεώρηση του πολιτικού προγράμματο. Θέλουμε να έχουμε και μια σαφή ανάλυση που θα ορίζει σαφείς προτεραιότητες, που θα ορίζει τα σημεία ε, στα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτερα, στα σημεία στα οποία υπάρχουν προβλήματα, στα σημεία ενδεχομένω που χρειάζεται να ορίσουμε ε, ω κοινοβούλιο διαφορετικέ προτεραιότητε. Τα ανώτατα επίπεδα, παραδείγματι, ορισμένων ε, κεφαλαίων. Χρειάζεται σοβαρή συνεργασία, σοβαρή δουλειά και ρωτώ η προσαρμογή των, της διοργανικής συμφωνίας πώς μπορεί να κλείσει όταν δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η διαμόρφωση της εξωτερικής υπηρεσίας. Όταν θα κρυθεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα υπόλοιπα που θα έχουμε να διευκρινίσουμε και που ενδεχομένως να πρέπει να κρυθούν ή να ενσωματωθούν καλύτερα από τη διοργανική ε, μέσα στα κεφάλαια για, την, για τις εξωτερικές σχέσεις. Αυτό δεν είναι τεχνική προσαρμογή της διοργανικής συμφωνίας. Ξεπερνά κατά πολύ την τεχνική προσαρμογή. Και γι' αυτό, Πρόεδρε, θα έλεγα, με τα λόγω γνώση, αλλά και σχετικά αυθόρμητα, ότι αποσύρω το έγγραφό μου. Αποσύρω το έγγραφο εργασίας και προτείνω και βέβαια την προσεχή εβδομάδα θα την αξιοποιήσω στο μέγιστο για να συζητήσω με τους ε, συντονιστές και τους λοιπούς συναδέλφους. Και προτείνω λοιπόν να εξαρτήσω την προσεχή μου δουλειά ε, από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ε, πολιτικό σχεδιασμό, για τη διοργανική συμφωνία και να ξεκινήσουμε προς τα τέλη Μαρτίου να ξαναβλέπουμε αυτή την υπόθεση με την προοπτική της ενσωμάτωσης της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής αναθεώρησης στην δουλειά αυτή. Γιατί αν δεν είναι τώρα η Επιτροπή σε θέση να αναλάβει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και να το ασκήσει, το έχω πει και εγώ νωρίτερα, θα το αναλάβουμε εμείς. Την πρωτοβουλία την αναλαμβάνουμε εμείς. Έχουμε εμείς το αίσθημα της ευθύνης αυτήν εδώ την Επιτροπή και θα το πράξουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ Ράιμερ για την πρόταση αυτή. Ο James Έλλης, έχει κάποιο σχόλιο και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. James. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πρέπει να εκφράσω την άποψη της ομάδας μου, γιατί τα άλλα μέλη της ομάδας μου δεν είναι παρόντα. Κάποιες παρατηρήσεις έχω ιστορικώς πως η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2000-2006 ε, είδαμε ότι περιείχονται αμφισημίες στις διατάξεις και σε αυτό το δημοσιονομικό κανονισμό υπάρχουν αμφισημίες 2009-2010 πάντα ήταν κάτι αμφίβολο όσον αφορά την προθεσμία και τους όρους διάμεσης αναθεώρησης, αλλά υπάρχει διαδικασία όσον αφορά την ανανέωση των δημοσιονομικών προοπτικών. Και έχω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ράιμερ. Τώρα θα συμβεί αυτό τα μέσα του 2011, διότι πλησιάζουμε ήδη διότι κάπως μας έχει γλιστήσει το χρονοδιάγραμμά μας. Το ερώτημά μου. Στις προτάσεις του Ράιμερ Μπέργκερ, στο έγγραφό του, που αφορά τη θέση που είχαμε στην Επιτροπή Προπολογισμών στην προηγούμενη θητεία που ακολουθούσαμε διαδικασία των τριών φάσεων και με την παράταση των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών δεν έχουμε δήλωση του Κοινοβουλίου ή αυτής της Επιτροπής Προπολογισμών για τη συγκεκριμένη άποψη. Θα ήταν χρήσιμο να υποβληθεί η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το καλοκαίρι, οι αρχέ του φθινοπόρου. Πούμε ποιε είναι οι δημοσιονομικέ προοπτικέ, ποια είναι τα αιτήματα τη Οικονομική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώ αντιμετωπίζετε αυτό και να επαναλάβω την άποψή μα ότι θα θέλαμε να έχουμε μια παράταση των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών. Διαφορετικά, ίσω κάπου χαθούμε στη συζήτηση. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα. Γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, ευχαριστώ, James. Πράγματι. Όπως λέει ο James, και ταιριάζει με αυτά που είπε και ο συγγητή μα. και αυτά που είπαν και άλλοι συντονιστέ. Πράγματι, η Επιτροπή Προπολογισμών, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ποια είναι η θέση του. Ποια είναι η θέση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εργασιών και λήψη αποφάσεων. Επί τη ουσία, ποια είναι η θέση του Budget Review και το νέο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, όπω προβλέπονται. Θα παρατείνουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές, ούτως ώστε στο μέλλον να συμπέσουν οι δημοσιονομικές προοπτικές με την θητεία του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή θα παραμείνουμε στην επταετία αυτού, το εξέτασε και η προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου και εμείς θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω. Σύμφωνα με το ωράριο να σταματήσουμε εδώ. Ευχαριστώ τους ε, εισηγητές στους ομιλητές. Ο Ράιμερ ανακοίνωσε το αποσύρει το έγγραφό του ότι θέλει να προσθέσει κάτι ο Ράιμερ. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στον τζέμι πολύ σύντομα. Αν θυμάμαι καλά, τη φιλόδοξη αυτή μεταρρύθ, ε, αναθεώρηση την έχουμε ε, ορίσει, την έχουμε ψηφίσει μάλλον στην Ολομέλεια με το ψήφισμα του συναδέλφου Σόγιαν και είχαμε συζητήσει εντατικά και εδώ μέσα στην Επιτροπή μας, αν δεν ναι. κάνω λάθος. Είχαμε βρει μάλιστα και συμβαστικές διατυπώσεις, όλα αυτά. Ε, εν πάση φαίνεται όμως ότι το Συμβούλιο και την Επιτροπή όλα αυτά δεν τα συγκινούν. Ελπίζω παρόλα αυτά να βρούμε μια ενδιαφέρουσα και σωστή πάνω απ' όλα εναλλακτική και να δούμε με την ησυχία μας το 2011, το 2012, πώς θα προχωρήσει η κατάσταση, πώς θα μπορέσει το Συμβούλιο να λύσει τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες. Ελπίζω όπως πάντα με μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Η Επιτροπή η, με την πρότασή της για τη νέα διοργανική συμφωνία μιλάει για την 1η Ιουλίου του 2011 όπου θα υποβάλει τις προτάσεις για, για ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή αναφέρεται αποκλειστικά στη μεσο, στην, ε, στο νέο πολιετή προγραμματισμό και καθόλου σε μία μέσο πρόθεσμη αναθεώρηση, την οποία εμείς περιμένουμε. Εμείς αυτό προσπαθούμε να ε, βάλουμε μέσα στην ε, συζήτηση. Με τις προτάσεις μας και με τις τροπολογίες μας βεβαίως θα πιέσουμε και θα ξεκινήσουμε τις πραγματεύσεις. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Από αυτά που μα είπε επιβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής, συγκρατούμε το εξή ότι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 11 Μαρτίου προβλέπεται η υιοθέτηση των νομικών κειμένων του Δημοσιονομικού Κανονισμού καθεστώς καταστατικό του προσωπικού και σε σχέση με τις εξωτερικές υπηρεσίες και αυτό θα ακολουθηθεί μερικές εβδομάδες αργότερα. Δεν έχουμε ισότερε λεπτομέρειε από το προσχέδιο θετικού προπολογισμού και χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών. 28 Απριλίου θετηθεί το σχέδιο προπολογισμού 2011 και το εγγράφο ως της Διοργανικής Συμφωνίας μήνα Μάιο. Το Σώμα θα θετήσει τις προτάσεις του όσον αφορά την τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, το budget review Ιούλιο-Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο το θέμα με το πολιτικό τίτλο ο ανεκτός, το ανεκτό επίπεδο σφαλμάτων, ο ανεκτός κίνδυνος σφαλμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να πάμε στο δεύτερο στάδιο των πρωινών μας εργασιών, δηλαδή τις ψηφοφορίες. Θα ζητήσω λοιπόν από όλους, καταρχάς από τους συντονιστές να διαπιστώσουν ότι πράγματι ότι είναι παρόντα όλα τα μέλη τους για να ψηφίσουν ή δεν έχουν τουλάχιστον παραπάνω από αυτούς ε, που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Επίσης ο καθένας σας ας έχει την κάρτα του διότι έχουμε αρκετές εκατοντάδες ψηφοφορίες. οι εκθέσεις που προτάθηκαν ε, οδήγησαν σε πολλές ε, φάνταστες προτάσεις και ε, τροπολογίες. Γκόραν, έχεις ερώτηση, όχι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την έκθεση της Συντόνια. Γκόραν, πρώτα απ' όλα έχω ένα σχόλιο. Ακόμα δεν λάβαμε όλες τις τροπολογίες στις γλώσσες που καταλαβαίνουμε. Πρόβλημα είναι αυτό, πραγματικά πρόβλημα. Αφορά και τις δύο εκθέσεις. 8 και 49 μας θέλει να νέα εκδοχή των τροπολογιών της εκθέσεως της Helga Triple. Μόνο γερμανικά κάποιες τροπολογίες και όχι στα αγγλικά. Και όχι στα σουηδικά, αυτό σίγουρο. Και αυτό ήταν πρόβλημα για όλες τις τροπολογίες της εκθέσεως ε, της ε, Συντόνια. Καταλαβαίνω. Έχει πιέσει και η γραμματεία της Επιτροπής Προπολογισμών και έχουν ε, πιέσει και μεταφραστές. Αλλά δεν είναι αποδεκτή η κατάσταση, είναι σημαντικότατη η ψηφοφορία. Και μάλιστα, όπως ακούσατε και στην προηγηθή σας συζήτηση, τους επόμενους μήνες θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό με το EAIS, με το προπολογισμό, την ενδιάμεση αναθεώρηση, τη διοργανική συμφωνία και θα έχουμε τεράστιες πιέσεις. Θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της μεταφράσεως, τη διαχείριση των προτάσεων, αλλιώ θα υπάρξει δημοκρατικό πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Και έχω ένα δεύτερο ερώτημα για την έκθεση για το GMES. σκιώδη συγητής μα η κυρία και η συγγήτριά μα, η Σκιώδη, μπορεί να τα εξηγήσει περαιτέρω. Έγιναν πολλέ διαπραγματεύσει με την Επιτροπή Ήτρε σχετικά με τα ποσά που θα προτείνουμε για, το πρόγραμμα, για το πρόγραμμα GMES. Το θέμα είναι ότι εδώ πραγματικά θα πρέπει να συζητήσουμε πώς σχετίζεται αυτός ο τομέας με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οπότε προτείνω να αναβληθεί το θέμα αυτό μέχρι την επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή μα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να συντονίσουμε τα ποσά με την Επιτροπή Ήτρε. Εφόσον η συγητή απουσιάζει, ίσω και γι' αυτό το λόγο θα ήταν χρήσιμο να γίνει κάτι τέτοιο. Ζητώ κύριε Πρόεδρε να αποφασίσετε κατά πόσο θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία επί τη εκθέσεω για το GMES. Πρόεδρο. ναι, ευχαριστώ Γκόχαν. Η κυρία Καβάριο και μετά η συντόνια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στον αφορά την αναβολή της εκθέσεως για το GMES, συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε και άλλους πόρους για το GMS e ε, και δεν διατίθενται στα πλαίσια του παρόντος προϋπολογισμού. Δεν υπάρχουν περιθώρια για τα χρήματα που χρειαζόμαστε για το GMS e Έχουμε στο 1α πολύ μικρά περιθώρια. Είναι σημαντικό όμως τις συζητήσεις για την αναθεώρηση αυτό να ληφθεί υπόψη. Όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης GMES, αλλά και για άλλες πολιτικές που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες συνθήκης της Λισαβόνας. Ταυτόχρονα όμως δεν θα πρέπει να αναβάλουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης, το GMES, γιατί είναι σημαντικό να αρχίσει αμέσως στην προβλεπόμενη περίοδο με τα προβλεπόμενα χρήματα και τα χρήματα που αναφέρονται στην έκθεση. Μια αναβολή όλων αυτών θα καθυστερήσει το πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικότατο για τους πολίτες, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, για το περιβάλλον, για τις φυσικές καταστροφές κλπ. Δεν συμφωνούμε λοιπόν. Και αν είναι να αναβάλουμε μόνο για δύο εβδομάδες μέχρι τις ψηφοφορίες στην Επιτροπή Ήτρε δεν λύνουμε τίποτα. Σε δύο εβδομάδες δεν θα βρούμε κι άλλους πόρους. Στην έκθεση ήδη συμπεριλαμβάνουμε τους μέγιστους ε, διαθέσιμους πόρους εντός των ισιουσών δημοσιονομικών προοπτικών. Δεν κερδίζουμε τίποτα με αναβολή και αν κινηθούμε κανονικά δεν υπονομεύουμε και τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Λοιπόν, καλό θα ήταν να μην αναβάλουμε. Έχω κάποιον που ζήτησε το λόγο. Δεν έχουμε χρόνο όμως για να συζητήσουμε επί της ουσίας. Την ουσία ούτε το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να ψηφίσουμε. Όσον αφορά το GMES, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Η αρμόδια επιτροπή είναι η επιτροπή Ήτρε. Θα ψηφίσει 18 του μηνό. Εμείς έχουμε συνεδρίες 17. Μπορούμε να ψηφίσουμε στι 17. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η Κομπίου να ψηφίσει πριν από την Ήτρε. Συμφωνείτε όλοι να κανονίσουμε να ψηφίσουμε πριν από την Ήτρε, αλλά για να δεχτούμε τα αίτημα σοσιαλιστών να μην ψηφίσουμε σήμερα. Σας ικανοποιεί αυτό, σας βολεύει, αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Επ' αυτού ζητήσατε το λόγο. Συντόνια. Πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, Πρόεδρε, θα ήθελα σας παρακαλώ να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Γιώργος Φάρμ. Ξεκινά πολύ καλά η ψηφοφορία. Συμφωνώ απόλυτα με τον σοσιαλδημοκράτη συνάδελφο, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστεί κανείς με μικτές γλωσσικές εκδοχές τροπολογιών για να καταλάβετε το ρυθμό των εργασιών από κάποια πράγματα και να κάνω και κάποια πρόταση. Έλαβα μεταφράσεις, επίσημες μεταφράσεις στα αγγλικά των τροπολογιών εχθές. Να μην μιλήσω τώρα για την πολωνική μετάφραση, διότι αυτό δεν είναι το στα όνειρά μου, δεν το περιμένω. Ηρωνεύομαι κάπως, αλλά δεν το περίμενα καν να γίνει αυτό για να καταλάβετε συνάδελφοι τι συνέπειες υπάρχουν πέραν από αυτές που ανέφερε ο Γιώραν. Εγώ που προετοιμάζω, ε, προετοιμάζω συμβιβασμούς επιγλωσσικών εκδοχών που δεν κατανοώ. Όπως σωστά είπατε κάποιοι από εσά και ήσατε σε επαφή μαζί μου και σας ευχαριστώ για αυτό, θεωρήσατε ότι δεν συμπεριέλαβα τους συμβιβασμούς σας. Κάποιοι από εσά βασισμένοι στην εξυπνάδα σας ε, θεωρήσατε ότι ε, έκανα διάκριση εναντίον σας διότι δεν συμπελεύα την τροπολογία σας και αναφέρω στους Ιταλούς συναδέλφους. Ήταν πολύ υπομονετικοί διότι κάθισαν και με βοήθησαν να καταλάβω, να μου εξηγήσουν τις τροπολογίες τους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεν αφορά μόνο τα Ιταλικά, αφορά όλες τις γλώσσες που δεν καταλαβαίνω εγώ και έχω επιλογή μεταξύ του να μάθω μια καινούρια γλώσσα, Ιταλικά, Ισπανικά, ακόμα το σκέφτομαι ποια θα μάθω. Αλλά στην πράξη τι σημαίνει. Ότι εγώ με τη μεγάλη υποστήριξη της γραμματείας που δεν είναι επαγγελματίες μεταφραστές οι άνθρωποι της γραμματείας άρα έχει και όρια αυτό που μπορούν να κάνουν. Λοιπόν μαζί με τη γραμματεία πρέπει να συνεργαστώ να προσπαθήσω να καταλάβω τις τροπολογίες να προσπαθήσω να τις καλύψω με συμβιβασμούς ε, με, ελήψη επισήμων μεταφράσεων και κάποιες τροπολογίε είναι τόσο συγκεκριμένε που μια αεραστεχνική μετάφραση ή μια διαστητική μετάφραση δεν λειτουργεί. Δεν ψάχνω να βρω δικαιολογίε, όχι, γιατί προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, αλλά έχουμε πρόβλημα, νομίζω. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ. Και όταν το γνωστοποίησα το πρόβλημα στη γραμματεία, μου είπαν ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που νόμιζα. Διότι, σύμφωνα με του κανόνε μα, η υπηρεσία μεταφραστική δεν έχει υποχρέωση να μας δώσει καμία μετάφραση του εγγράφου διότι δεν τηρούμε τις προθεσμίες. Έπρεπε να υποβάλουμε τις προτάσεις δύο-τρεις εβδομάδες πριν νομίζω. Οπότε, για τις εργασίες μας αυτή είναι, τι να σας πω, είναι κάτι απίθανο. Και δεν μιλάμε και για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, τεράστια κείμενα, μερικές φράσεις, δύο σελίδες είναι το κείμενο. Γιατί αναφέρθηκα εκτενώς αυτό, διότι θα ήθελα το μήνυμα να διαβιβαστεί στους υπευθύνου του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να καταλάβουν τι συνέπειες έχει αυτή η κατάσταση για τη δουλειά μας και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα που επικρατεί στην μεταφραστική υπηρεσία. Δεν φταίω εγώ, αλλά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από εσά που λάβατε τις συμβαστικές προτάσεις πολύ αργά για να μπορέσετε να τις επεξεργαστείτε αλλά θα έπρεπε να τις προετοιμάσω μόνο χθες το βράδυ θα μπορούσα να τις προετοιμάσω διότι μόλις χθες ε, μπόρεσα να καταλάβω τις διάφορες προτάσεις χρησιμοποίησαμε τα διαθέσιμα εργαλεία βλέπετε συμφωνώ και πάλι με τον Γιώραν και πιστεύω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα. Δεν ξέρω να έχουμε κάποιες προτεραιότητες, να εξετάσουμε τι γίνεται με τη μεταφραστική υπηρεσία. Δηλαδή η δομή της μεταφραστικής υπηρεσίας θα πρέπει κάπως να προσαρμοστεί για να μπορεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα των εργασιών μας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Προτείνω να σταματήσουμε εδώ με αυτά τα προβλήματα. Τίθεται πρόβλημα ουσιαστικό βέβαια που αφορά και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουμε το δικό μας χρονοδιάγραμμα εργασιών σε περίπτωση των συνεδριάσεων των συντονιστών και τις προθεσμίες που καθορίζει ο ίδιος ο εισηγητής. Όσο έχουμε καθυστέρησης ανάντι, εμπλέκονται και σταματούν οι εργασίες κατάντι. Λοιπόν, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Το ΕΛΚ έχει δικαίωμα 16 ψήφων και μου λένε ότι τα 16 μέλη του ΕΛΚ είναι εδώ συμπεριλαμβανομένου εμού του ιδίου Δηλαδή, αν φτάσει η η θα ψηφίσω, αλλά προειδοποιήστε με. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες έχουν 11 ψήφου, οι άλλοι 5, οι πράσινοι 3, οι συντηρητικοί 3, η Γκουε 2. Σας τα θυμίζω αυτά, έτσι. Η κυρία Καρβάγιο. Πρόεδρε, λυπούμε. Θα ήθελα απλώ να διευκρινίσω το GMS, ποια είναι η τελική απόφαση. Θα το αναβάλουμε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης. Εάν αποφασίσουμε μια μέρα πριν από την Ήτρε, από την Επιτροπή Μηχανίας, χάνουμε και τη διαπραγματευτική μας ισχύ. γιατί είναι πιο κοντά στην Επιτροπή Ήτρε. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Καλύτερα, όχι μια μέρα μόλις πριν από την Ήτρε, αλλά βέβαια εσείς κρίνετε. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Σας αντιλαμβάνομαι. Όμως η απόφαση ελήφθη. Σημαντικό είναι στις διαπραγματεύσεις με την ΙΤΡΕ ο εισηγητής μας, ο κ. Σαββάτ, ο οποίος ε, έχει αυτές τις διαπραγματεύσεις, να τις διεξαγάγει όπως πρέπει και σε συνεννόηση με τους συντονιστές. Κύριε Άλβαρο, εσείς πολύ γρήγορα. Ναι, Πρόεδρε, έχω το εξή μόνο. Προθεσμίες που πρέπει, που θα έπρεπε να έχουν τηρηθεί. Αφού χτε λάβαμε μόλι τα τελευταία, τις τελευταίες εκδόσεις, δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για προφορικές τροπολογίες, ούτε για χωριστέ ψηφοφορίες. Και ω εκ τούτου θα θέλαμε ω ομάδα να επισημάνουμε κάποια σημεία στα οποία θα θέλαμε να δώσουμε προσοχή. Δεν ξέρω ε, όμως ακριβώς ποια είναι η διαδικασία, γιατί όταν έχουμε προθεσμίες για προφορικές τροπολογίες είναι διαφορετικές ίσως από την, ε, την προθεσμία για το αίτημα ε, να ψηφιστεί σε τμήματα η τροπολογία. Ποια είναι η κατάσταση, Πρόεδρε, ο Πρόεδρος. Αγαπητέ φίλε, μη φοβήστε. Θα είμαι πολύ πολύ ευέλικτος στην υπόθεση αυτή, διότι πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει η απόφαση που θα ληφθεί από την Επιτροπή των Προπολογισμών να ληφθεί με τα λόγω γνώση και να αντιστοιχεί στα πολιτικά κριτήρια με την σαφή και ευγενή έννοια του όρου. Δηλαδή με απόλυτο σεβασμό του κανονισμού. Τώρα, εάν για λόγους προθεσμιών ή άλλους η κατάσταση είναι τέτοια που θα χρειαστεί να ερμηνεύσουμε ευέλικτα, αν θέλετε, τον κανονισμό για να εξασφαλίσουμε το επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα, θα το πράξουμε. Και με αυτή την ε, ε, ενθάρρυνση και τις προσχέσεις για ευελιξία προτείνω να ξεκινήσουμε την έκθεση της Χέλγα αφού έχει λιγότερες τροπολογίες από αυτήν τη συντόνια. Σας παραπέμπω λοιπόν στους καταλόγους των τροπολογιών σας και στην κάρτα για την ψηφοφορία. Ποιος δεν έχει κατάλογο ε, ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ. Κοιτάξτε να σας πω το ΕΛΚ έχει τον επικεφαλή του, έτσι. Ποιος είναι. Α, διανέμεται. Ωραία. Διανέμεται λοιπόν η Έλγα. Η έκθεση τη Έλγα. σου ψηφοφοριών. Bon, ça y est, le PPE est en état de voter. Είμαστε έτοιμοι, ΕΛΚ. E, Ξεκινώ. Τροπολογία υπαριθμών 1. Utah Χάουκ. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 2 του κυρίου Βον. Μετά την ε, τέταρτη παράγραφο λέει ο πρόεδρος. Υπέρ είναι η συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία θα κάνουμε μόνο αν βλέπω ότι δεν ε, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παράγραφο 3, Φερνάντς Καρίγα, προφορική τροπολογία εδώ, μέτρο προφορική τροπολογία, τη εισηγητρίας που προσθέτει τη φράση και να αναθεωρηθεί αναλόγως στον άτοτο όριο. Υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές αλλά στη ψηφία, εγκρίνεται ε, τρεις τροπολογίες των υπαριθμών 5 παράγραφο. Έχουμε τη συμβαστική υπαριθμών 1 καταρχάς, η οποία θα αντικαταστήσει την 4 του κυρίου Χάγκλουντ. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής. Αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η 4, αλλά δεν καταπίπτει η 6, δεν καλύπτεται. Την 6 της κυρίας Βέρτμαν, η συγγετρία είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ, ευχαριστώ κατά. Ουδής. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 του κυρίου Πόρτας, η συγγετρία δεν την βρίσκει καλή. Υπέρ, κύριος Πόρτας μόνο και άλλος ένας. Κατά. Όλοι οι άλλοι. Κύριε Πόρτας, ατυχία. Απορρίπτεται. Βον και Φέρμ υπαριθμών 7 δεν τις συμπαθεί η συγκίτρια της τροπολογίας. Αυτές υπέρ. Οι σοσιαλιστές και η κυρία εκεί. Κατά η πλειοψηφία απορρίπτεται. Στην παράγραφο 7. Τροπολογία Φερνάντες Γκαρίγα με προφορική τροπολογία με τον όρο θεσμός θεσμό Η συγγετρία είναι υπέρ. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο, κάτι ξέχασα. Κάτι ξέχασα. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο, γυρνάμε πίσω. Ξέχασα την 8 του κύριου Πόρτα, όπου η συγγήτρια είναι υπέρ αυτή τη φορά. Υπέρ, παρακαλώ. Πλειοψηφία. Κατά. Μια ψηφία Αποχέ. Εγκρίνεται. Μπράβο, κύριε Πόρτα. Παρηγορηθείτε. Στην 9 τώρα. Έχουμε μια μικρή προφορική τροπολογία με το θεσμικό όργανο της συγκήτριας. Ε, υπέρ, η συγκήτρια είναι υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Κύριε Βόν, στην τροπολογία 10, Πρόεδρε, η συγκήτρια ζητεί να γίνει ψηφορία σε τμήματα από ό,τι κατάλαβα. ενδέχεται το πρόβλημα είναι μάλλον γλωσσικό. Εμείς προσπαθούμε ως ομάδα να ενημερώνουμε όσο δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να διαγράψουμε τις δύο λέξεις how much of, τρεις λέξεις, πόσο από ή σε ποιο βαθμό. Ελπίζω αυτό να είναι αποδεκτό για την εισηγήτρια. Ως προφορική τροπολογία. Η εισηγήτρια τι λέει. Ναι, λέει η κυρία Τρίπελ, συμφωνώ. Συμφωνεί λοιπόν η συγγήτρια και ο εκ τούτου και ο Γκέραν. Το σύνολο της τροπολογίας ε, με την τροποποίηση αυτή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Βόν. Στην 11 πάλι του κύριου Βόν, υπέρ κατά η Μπάρμπαρα. Μα τι είναι αυτό τώρα, Μπάρμπαρα, έχεις, ε, κάτι δικό σου με τον κύριο Βόν, τα έχεις βάλει μαζί του τώρα, τέλος πάντων δική σου υπόθεση. Παρά τη στεναρή <laughs> αντίσταση της Μπάρμπαρα κρίνεται η τροπολογία και πάμε στον κύριο Μάνκα στη 12, δηλαδή η συγγήτρια είναι κατά της τροπολογίας, υπάρει παρακαλώ. Αχα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. η ομάδα μου να μου πει αν ψηφίζουμε υπέρ ή κατά. Όλοι είμαστε υπέρ λοιπόν, εκτός της ε, εισηγήτριας. Άρχιτη ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 6 κατά. Κύριε Μάνκα, πιστεύω να είστε ικανοποιημένο, να είναι μάλλον ικανοποιημένο ο κύριο Μάνκα. Στη 13 Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Η πλειοψηφία είναι υπέρ της συμβαστικής και ως εκ τούτου αντικαθίσταται η 13 από τη συμβαστική. Ε, τώρα, να πάλι ο κύριος Βον, ο οποίος φανταζόμαστε ότι καλύπτεται από τη συμβαστική 2, έτσι. Μάλιστα. Πολύ καλά. Και προχωρούμε στο, στην τροπολογία 15 που έχει μια συμβαστική υπαριθμών 3 της εισηγητρίας. Υπέρ παρακαλώ της συμβαστικής 3. Ευχαριστώ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται, αντικαθιστά λοιπόν τη 15 και ταυτόχρονα καλύπτει και την 16. Έτσι δεν είναι, Φερνάντης και καρύγα. Πάμε στη 17, τον κύριο Πόρτας, όπου τώρα δεν ε, ε, είναι υπέρ η συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Αχα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Και άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ παρακαλώ, ναι. Πέρας της ψηφοφορίας, τι λέει το μηχάνημα. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 23 ψήφικα κατά. Κύριε Γκρέσλε. Θα ήθελα, Πρόεδρε, εδώ στην τροπολογία 18 να στήσω ψηφοφορία σε, δύο, σε τμήματα. Είχαμε καταθέσει το αίτημα σχετικά αργά, αλλά έχει εδώ τη θέση του στην προσθήκη του κύριου Πόρτας. Δηλαδή, μέχρι εκεί που λέει «which is already stretched» και μετά θεωρεί ότι «considers that the market» κτλ. χωριστά ως δεύτερο τμήμα. Καταλάβατε όλοι, λέει ο πρόεδρος. Κόβουμε στο which is already stretched. Στο πρώτο αυτό τμήμα λοιπόν, η συγκίτρια τι λέει. Κατά, πρόεδρε. Κατά. Καλώς, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά πρώτο Στο δεύτερο τμήμα η εισηγήτρια πάλι είναι κατά. Κύριε Φερνάντσου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στόχος είναι να διατηρήσουμε το πρώτο τμήμα, να αποσύρουμε το δεύτερο να αποσυρθεί μάλλον το δεύτερο και να υπερψηφίσουμε το τελευταίο τμήμα. Λέει ο κύριο Φερνάντς. Je parle de l'amendement original. Όχι, όχι, εγώ είμαι στην αρχική διατύπωση, στην αρχική τροπολογία. Ένα λεπτό, λέει ο πρόεδρος, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η τροπολογία του κυρίου Φόρτας έχει σαν στόχο όχι... Φερνάντες μάλλον θέλει ο πρόεδρος όχι να αντικαταστήσει την τροπολογία 11. Όχι να διαγράψω θέλω λέει ο κύριος Φερνάντης. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, εγώ κατάλαβα λάθος. Ο κύριος Πόρτας θέλει να αντικαταστήσει την 11η ε, παράγραφο με την τροπολογία 18. Ζητήθηκε το, η ψηφοφορία σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα απερίφθη της 18. Ένα λεπτό να δούμε και το δεύτερο τμήμα τώρα. Ε, κυρία Τρίπλ, πρόεδρε, πρέπει να ξαναψηφίσουμε ε, γιατί από ό,τι κατάλαβα εγώ το ΕΛΚ δεν ψήφισε όπως σκόπευε να ψηφίσει ή όπως είχε προεξαγγείλει ότι θα ψηφίσει. ειναι καλά κατάλαβε η ΕΛΚΑ. Κυρία Γκρέσλη, πρόεδρε, εγώ νόμιζα ότι ψηφίσαμε μόνο την προσθήκη του κυρίου Πόρτας και όχι το αρχικό κείμενο. Για την προσθήκη είμαστε κατά του πρώτου τμήματος της προσθήκης του κυρίου, του Πόρτας. Αλλά τα θεσόμεθα υπέρ του δεύτερου τμήματος της προσθήκης του κυρίου Πόρτας που είναι άλλωστε το αρχικό κείμενο. Κοιτάξτε, λίγο, ο ένα λεπτό. Εγώ σα καταλαβαίνω, ο κύριο Πόρτα είναι εδώ, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι προσθήκη, αλλά αντικατάσταση η τροπολογία του. Για την ακρίβεια είναι διαγραφή. Θέλει να απαλείψει ένα μέρος του κειμένου. Άρα, εάν απορρίψουμε την τροπολογία του κυρίου Πόρτας, έχουμε αυτόματα υιοθετήσει την 11η παράγραφο.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 Alors, recommençons. Moi, je, je n'y comprends rien. Euh, je... δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Ας ξαναρχίσουμε λοιπόν. Μου, ζητάτε το μηδέν να το χωρίσω στα δύο και να ψηφίσω δύο τμήματα του, του μηδενός. Του τίποτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κύριε Φερνάντος, για εξηγήστε λίγο τι θέλετε. Πρόεδρε, είναι πιο απλό εάν πάρουμε το αρχικό κείμενο Τώρα για του ε, κανονισμού, δεν ξέρω τι ισχύει, ποιο άρθρο και πώ θα το κάνουμε κτλ. Αλλά αυτό που θέλουμε εμεί είναι το εξή. ότι συμφωνούμε με το πρώτο τμήμα, ενώ για το δεύτερο θέλουμε να το καταργήσουμε. Και συμφωνούμε και για το τρίτο τμήμα. Τώρα αν μας πάτε σε τροπολογία πόρτας που θέλει να διαγράψει όλο το, δεύτερο μισό, τότε τι να σας πω, δεν βγαίνει άκρη, πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε με βάση το αρχικό κείμενο. Non. Bon. Alors voilà ce que je vous propose. Quelle histoire. Il y a trop de portugais dans cette histoire. Bon, alors, traduire en, en polonais, vous voulez consentir. Bon. Ας δούμε λοιπόν από εδώ και προς τι γίνεται. Ψηφίζω την τροπολογία του κ. Πόρτας, που είναι πιο μακριά από το αρχικό κείμενο. και που ζητεί να καταργηθεί το δεύτερο τμήμα ολόκληρο της παραγράφου. Θα δούμε μετά την ψηφορία σε τμήματα. Λοιπόν, πρώτον, για την τροπολογία πόρτας μόνο, χωρίς ψηφορία σε τμήματα, όλο το, όλη την τροπολογία. Η συγκεκριμένη είναι κατά. Καλώς. Κατά. Όλοι λυπή. Συνεχίζω να βρούμε μια διαφορετική λύση τώρα περιμένετε. Θα κάνουμε το εξή. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Σε τμήματα δηλαδή θα ψηφίσουμε όχι την τροπολογία πόρτας, αλλά το ίμιση της δεύτερης φράσης της παραγράφου, της 11 της τροπολογίας 18, της μάλλον παραγράφου 11. Δηλαδή κόβω το κείμενο πάω στο underlines especially, εκεί που είναι οι παχείς λιπαροί χαρακτήρες, ιδιαίτερα υπογραμμίζει ότι αν πρόσθετοι βοηθοί προσληφθούν στις Βρυξέλλες, ε, αυτό θα έχει επιπτώσεις προς τον, ε, το χώρο για γραφεία κτλ, που ήδη είναι προβληματικός. Ποιος θέλει το κείμενο αυτό να μπει μέσα στο ψήφισμά μας. Να μείνει μέσα στο ψήφισμα. Πρέπει να μείνει μέσα στο ψήφισμα. Ποιος είναι υπέρ. Μένει μέσα στο ψήφισμα. Καλώς, ας κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Δηλαδή το ΕΛΚ από ό,τι φαίνεται θέλει να διαγραφεί αυτό το κείμενο. Αλλά άλλοι θέλουν να το διατηρήσουν. Καλώς, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Μεγάλο suspense. 18 υπέρ, 18 κατά. Δεν είναι τροπολογία, είναι αρχικό κείμενο, δεν διαγράφεται. Μένει το κείμενο μέσα στην περίπτωση ψηφία. Τώρα, δεύτερο και τελευταίο τμήμα θεωρεί ότι η παρουσίαση το Μάρτιο της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια στους τρεις τόπους εργασίας είναι ε, ουσιώδεστατες σημασίες. που θέλει να παραμένει το κείμενο αυτό. Όλοι ναι. Συμφωνούμε. Κατά ουδείς αποχές. Άρα, μετά από όλη αυτή την ιστορία, παραμένει η ενδεκάτη παράγραφος όπως την είχε αρχικά διατυπώσει η συγκεκριά. Ωραία. Υδρώσαμε, όλα τα καταφέραμε. Παράγραφος 18 ήταν αυτή, η τροπολογία 18 μάλλον. Πάμε στην τροπολογία 19 με ένα δεύτερο τμήμα το οποίο καταπίπτει αν εγκριθεί 18. Η 18 έχει εγκριθεί λέει ο πρόεδρος. Α, όχι δεν εγκρίθηκε. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε τη 19. Η συγγετρία είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής. Υπέρ παρακαλώ. Le vote... Και πάλι ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτε η ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρασε 19 υπέρ, 15 κατά εκκρίνεται. Και περνούμε στην τροπολογία της Ίνγκε Γκρέσλε την 20. Δεν πέρασε 18, άρα δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Και πάμε σε, στο τμήμα αυτό, σε δύο τμήματα, με το και ή Στρασβούργο. Την αποσύρω, Πρόεδρε, λέει η κυρία Γκρέσλε. Αποσύρεται λοιπόν και άρα δεν θα κάνουμε ψηφορία για την υγιεινή των χειρών στο χώρο εργασίας πολύ καλά. Ε, μια τροπολογία από την Ιβυρική Χερσόνησο, Φερνάντας Γαρίγα, 21, υπέρ παρακαλώ, κατά εγκρίνεται. Ας πάμε στην 22 που είναι μάλλον βαβαρέζικη, η συγγήτρια είναι υπέρ, οι άλλοι είναι όλοι υπέρ, υπάρχει κανείς κατά, όχι εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην κυρία Χολμαϊρ. Ο κύριο Βόγκαν που είναι πολύ δραστήριο τροπολογία 23 είναι υπέρ ο εισηγητή. και υπέρ είναι το ΕΛΚ και άλλε ομάδε. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν. Ξαναβρίσκουμε. Ο κύριο Πόρτα κατέπεσε στην 24. Όμω δεν καταπίπτει στην 25. 25 κύριο Πόρτα, είναι αρνητικό ηγητή. Ποιο είναι υπέρ κατά πλειοψηφία απορρίπτεται 26 Φερνάνδες και Καρίγα εισηγητής υπέρ αν αποτελεί προσθήκη κύριε Φερνάνδες ευχαριστώ έχω προφορική τροπολογία που αντικαθιστά το αρχικό κείμενο όπου λέει να επιδιωχθεί πιο αποτελεσματική επαγγελματική πολιτική όσον αφορά τις βαθμίδες, να αντικατασταθεί αυτό αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και προσθέτουμε και επαγγελματική πολιτική για το προσωπικό. Αποτελεσματική διαχείριση λοιπόν ανθρωπίνων πόρων εν τέλει και επαγγελματική πολιτική για το προσωπικό. αυτήν τελική εκδοχή. Έτσι το ερμήνευα και εγώ. Θεωρούσα ότι πρόκειται περί προσθήκης και όχι περί αντικαταστάσεως. Εμπλουτίζεται το κείμενο και συγκητής είναι υπέρ. Υπέρ ποιος είναι, υπέρ της τροπολογίας, όσο τροποποιήθη προφορικός κατά. Αποχές εγκρίνεται υπό αυτή τη μορφή. Φτάνουμε στην 27. Εκεί υπάρχει μια ψηφοφορία κατά τμήματα. Έχουμε Cost and Energy Efficient Buildings Policy. Το πρώτο τμήμα, εισηγητής είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Η πλειοψηφία κατά. Εν συνεχεία, δεύτερο τμήμα. Including with regard to location. Εδώ έχουμε suspense, διότι έχει ελεύθερη ψηφό το ΕΛΚ. είναι κατά. Λοιπόν, πάμε ηλεκτρονικά, ξεκινάμε. Including with regard to location. Και το ΕΛΚ είναι κατά. Ξεκινάει η ψηφοφορία, τελειώνει η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ νίκησε 17-15. Λοιπόν, 28. Η Ίγκε που την υποστηρίζει η ΕΛΚΑ. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Ε, κατά. Ψηφία υπέρ. Η Ίγκε νικά. 29. Βόγκαν. Αποσύρεται. 30. Βόγκαν. Αντικαθίσταται από συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ τη συμβαστική 4. Κατά. Αντικαθιστά λοιπόν την, την τροπολογία 30, τη συμβαστική. Και καλύπτει αρκετές τροπολογίες από ό,τι μου λέγουν. Για την 31 η πρώτη φράση καλύπτεται από προηγηθήσεις παραγράφους, το δεύτερο τμήμα καλύπτεται από τη ψηφοφορία για τη συμβαστική 4, οπότε ψηφίζουμε μόνο το τελευταίο τμήμα που αφορά το The House of European History. Είναι υπέρ, συγκεκριτής ποιος είναι υπέρ. Χαμογελάω, Σαλβαδόρ, δεν ξέρω γιατί, κατά. Ουδείς αποχές. Καμία αποχή. Λοιπόν, ε, χαίρεται πολύ ο Σαλβαδόρ και πάμε στη Γιούτα, στην 32. Συγητής εναντίον, υπέρ της 32. Κατά. Δεν ψηφίζουν πολύ. Αποχές. Νομίζω ότι περισσότεροι είναι εναντίον, ε. Κάποιοι σοσιαλιστές ψήφισαν υπέρ. 33 μάνκα που αντικαθίσταται από τη συμβαστική 5. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής προτάσεως 5. Κατά. Σημειοψηφίε σοσιαλιστές εγκρίνονται. 34 μάνκα. Συγητής κατά. Ποιος είναι υπέρ της 34 μάνκα. κατά απορρίπτεται 35 Χολμάιερ καλύπτεται από τη συμβαστική 4 ψηφίζουμε το τοροποιημένο σχέδιο εκθέσεως ποιος είναι κατά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια λοιπόν στην ΕΛΓΑ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που ψήφισαν με αποτελεσματικό τρόπο σε λογικά όρια μπορούμε να περάσουμε στην έκθεση της Συντόνια Λουκιεύσκα. Και έχουμε 200 τροπολογίες εδώ. Όχι, 118, 118. Λοιπόν, υπάρχει πρόταση συντόνια, τη συντόνια να ψηφίσουμε πρώτα τις συμβαστικές τροπολογίες. Μαζί. Όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Κάθε μία ξεχωριστά. Αυτό τι σημαίνει. Ότι θα ψηφίσουμε αρχικά όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, όχι με τη σειρά που ε, καταφθάνουν. Oui, dans l'ordre alphabétique. Mais je veux dire, euh, je commence par le... Ξεκινάμε τη συμβαστική Α, πάμε μετά στη Β και μετά θα επανέλθουμε στις ενδιάμεσες ψηφοφορίες. Περί αυτού πρόκειται, καταλάβατε. Όλοι έχετε λοιπόν το κείμενο των συμβαστικών τροπολογιών σε μια γλώσσα που καταλαβαίνετε, έτσι. Ο καθένας από σας καταλαβαίνει. Εάν χρειάζονται εξηγήσεις θα δοθούν. Ξεκινάω λοιπόν από τη συμβαστική Α. Γκόραν. Λυπάμαι, Πρόεδρε, που σας ε, διαταράσω ευθύ εξ αρχής την ψηφοφορία, αλλά αυτή η τροπολογία που αφορά το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως, όταν συζητήσαμε το θέμα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγγραφο του Χάιμερ Μπέργκε. θα ήθελα να ζητήσω από την συγγήτρια μήπως θα μπορούσαμε να, να συμπεριλάβουμε κάποιο προσδιορισμό για τον χρονισμό, διότι εδώ ζητάμε μια πρόταση για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Θα ήθελα να συμπεριλάβουμε τη φράση που είχαμε στη συζήτηση με τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι, δηλαδή να ζητήσουμε πρόταση πριν το τέλος του πρώτου εξαμήνου 2010. Αυτό προτείνω εγώ. Πρόεδρος, πρόκειται περί προφορικής τροπολογίας, προτάσεως για προφορική τροπολογία της εισηγήτρες, που συμφωνεί η εισηγήτρια βεβαίως. Ευχαριστώ Γκόραν, ευχαριστώ Συντόνια Ψηφίζουμε λοιπόν τη, συμβαστική τροπολογία α κεφαλαίο λατινικό με τη διευκρίνηση για το χρονοδιάγραμμα, για το πρώτο εξάμεινο. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ σας. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη βαστική Β της εισηγήτριας. Υπέρ. Α, όχι, συγγνώμη. Ο κύριος Αλβάρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν ήταν τυχαίο που ρώτησα νωρίτερα αν θα μπορούσαμε να έχουμε ευελιξία προς τις προφορικές τροπολογίες. Ε, καταρχάς βλέπω στο αγγλικό κείμενο ένα λάθος γλωσσικό. Το which μεταξύ του ability και του is. Αλλά αυτό είναι μάλλον ζήτημα που μπορούν να διορθώσουν οι γλωσσομαθείς. Αλλά θα ήθελα να πω το points out the use και να προσθέσουμε and education και εκπαίδευση. Όχι μόνο δηλαδή τη νεολαία, αλλά τη νεολαία με την εκπαίδευση της. Δεν αρκεί να μιλήσουμε μόνο για νεολαία. Θα ήθελα να βάλουμε και την εκπαίδευση μετά τη λέξη youth. Κυρία Συγήτρια, από ό,τι κατάλαβα, αναφέρεται στη δεύτερη αναφορά της νεολαίας στη συμβαστική Β. Αν περί αυτού πρόκειται, συμφωνώ, αλλά όχι στην πρώτη αναφορά στη νεολαία, youth. Από ό,τι κατάλαβα θα λέει το κείμενο. Υπενθυμίζει ότι η επένδυση στη νεολαία και στην παιδεία σημαίνει επένδυση στο σήμερα και στο μέλλον. Τότε συμφωνώ, αν περί αυτού πρόκειται. Ναι, youth and education, ναι. Ο κύριο Αλβάρο λέει ότι δεν είναι αξία η νεό, της νεολαία. Το λέει αυτό γιατί είναι νέος. Αυτό μα τα λέει έτσι. Λοιπόν, με αυτέ τι διευκρινήσει, αυτή τη σημαντική διευκρίνηση, τον ευχαριστούμε για αυτό. Ποιο είναι υπέρ τη σημαστική τροπολογίας Β κεφαλαίο. Κατά. Αποχές ομόφωνη έγκριση. Πάμε στην σε λατινικό συμβαστική. Ποιο δεν υπάρχει ανάγκη εξηγήσει, όλα είναι ξεκάθαρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική τροπολογία δι λατινικό της ηγήτριας. Εκεί ζήτησε ο Γκόραν να πει κάτι. Ναι θα ήθελα να ζητήσω όταν μιλάμε για και... Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Αργότερα θέλω να κάνω αυτή την πρόταση. Καλώς. Όσον αφορά το κεφαλαίο D, λατινικό, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική ε. Συντόνια. Έχω σημαντικό σχόλιο που αφορά τη συμβαστική ε. Η τροπολογία 27 δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμβαστική. Άρα θα πρέπει να ψηφιστεί όταν θα ψηφίσουμε κάθε τροπολογία ξεχωριστά. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση συντόνια, λέει ο Πρόεδρος. Δεν αλλάζει το κείμενο συμβαστική ε, όμω θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η συμβαστική δεν συμπεριλαμβάνει υπόψη την τροπολογία 27. Λαμβάνει υπόψη άλλε τροπολογίε, αλλά όχι την 27. Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Το ΕΛΚ έχει κουρασμένο χέρι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα συμβαστική F λατινικό. Συμβαστική F Α, βλέπω κακές προθέσει εδώ. Ο κ. Αλβάρο ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ ζητούμε την χωριστή σε τμήματα ψηφοφορία. Στο δεύτερη παράγραφο, εκεί που έχει αλλάξει το more substance και το especially in the field of climate change, environment and social policies θέλουμε να διαγραφεί αυτό να ξαναμείνουμε στο αρχικό κείμενο της δεύτερης, του δεύτερου της παραγράφου αυτής. Donc vous demandez ζητάτε κατά τμήματα ψηφοφορία. Κάνουμε διάκριση μεταξύ ενός πρώτου τμήματο που δεν λαμβάνει η υπόψη το climate change κλιματική αλλαγή και δεύτερο τμήμα που λαμβάνει υπόψη την φράση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Περί αυτού πρόκειται, όχι. Όχι, να το πω αλλιώς. Αυτή η δεύτερη τροποποίηση που αφορά την, το περιβάλλον και τις κοινωνικές πολιτικές θέλουμε να διαγραφεί, ώστε να επανέλθουμε στο αρχικό κείμενο. Αυτό που λέει with substance and resources δηλαδή στο αρχικό κείμενο, χωρίς εξειδίκευση ως προς τους πόρους θυμάστε τη συζήτηση την οποία είχαμε διεξαγάγει και πριν από τα Χριστούγεννα, ότι δεν ήταν σαφέ ε, το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένου τομεί ε, με δεδομένη τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση κτλ. Μάλιστα. Ορίστε, James. Euh, να προτείνω να ψηφίσουμε 43 και 44 ξεχωριστά. Διότι συμφωνώ με τον κύριο Αλβάρο τελικά. Αυτό που έλεγε το αρχικό κείμενο το 43 είναι αυτό που αφορά το 2020. Είναι απλούστο να αποσυρθεί η συμβαστική τροπολογία και να ψηφίσουμε τις 43 και 44, λέει ο Πρόεδρος. Όχι. Δεν ξέρω τι ζητάει συντόνια. Πέστε μας συντόνια, πώς θέλετε να ψηφίσουμε. Κοιτάξτε, προ... προτείνω να ψηφίσουμε ξεχωριστά στον φασιβαστική τροπολογία. Δεν συμφωνώ όμως να απορριφθεί η συμβαστική τροπολογία διότι περιέχει στοιχεία από τροπολογίες που δεν είναι καν από την ομάδα μου. Οπότε θα ήταν κατά των ε, συμφωνιών των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν. Πρόεδρο, εν τη αυτή περιπτώσει ψηφίσαμε, θα ψηφίσουμε μάλλον το πρώτο τμήμα τη τροπολογία. Welcomes the Commission's ε, working ε, document on the Commission's 2020 strategy που δείχνει ποιε κατευθύνσει θα ακολουθήσει στο μέλλον αντιμετωπίσει πραγματικέ προκλήσει που χρειάζεται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βάσει αυτή τη γενική συζητήσεω για, για την οικονομική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύει ότι αυτή η στατική θα πρέπει να τονίζει περισσότερο κλπ. κλπ. και σταματάμε στο more substance. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το πρώτο τμήμα τη σημαστική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 13 ψήφοι κατά. Οπότε αυτό το τμήμα εγκρίνεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα τώρα. with more substance, especially in the field of climate change, environment and social policies. Αυτό που δεν θέλει ο κύριος Αλβάρο. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Η φιλελεύθερη και συντηρητική είναι στη μειοψηφία, οπότε εγκρίνεται και αυτό το τμήμα. Πάμε τώρα στη συμβαστική G λατινικό της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Α, η εισηγήτρια να πάρει το λόγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Έχω ένα σχόλιο προφορική τροπολογία που αφορά τη συμβαστική G λατινικό, τη προφορική μου τροπολογία, διότι κάτι συνέβη στο γραφείο υποβολή των εγγράφων και σοσιαλι... ένα στοιχείο των σοσιαλιστών αρχικής τροπολογίας που δεν παρατήρησα έβαλαν τη λέξη traditional, παραδοσιακή, και δεν το είδαν, δεν είχε υπογραμμιστεί στο έγγραφο. Εν τι αυτή περιπτώσει, σημειώνω την αντίρρηση που υπάρχει για τη λέξη traditional και η προφορική μου τροπολογία αντικαταστεί το traditional με fundamental. Έχετε και το κείμενο. Και το δεύτερο, η δεύτερη προφορική τροπολογία, τρίτη γραμμή, λέει ο πρόεδρος. Το traditional στη τρίτη γραμμή. Και μετά έχω προστίκη όσον αφορά τη συμβαστική G λατινικό, μετά τον οριζόντιο χαρακτήρα, horizontal character, να προσθέσουμε την εξής φράση Σας ευχαριστώ κύριος Αλβάρο. Ευχαριστώ πολύ για να διευκολύνω την κατάσταση θα μιλήσω αγγλικά. Η ομάδα μου θα υποστήριζε το G, το λατινικό. Έχουμε ένα πρόβλημα με ένα κομμάτι. Μέσω προφορικής τροπολογής επιληθεί. Το Common Agriculture να διαγραφεί. Χρησιμοποιούμε πόρους από το κονδύλι για τη Γεωργία, για την Ευεζωνική στην Ήπεθρο, για το Γαλιλαίος αν θέλετε το πείτε ρητά ότι δεν μπορούμε να πειράξουμε αυτά τα κονδύλια, εντάξει, αλλά θα πρέπει να επηρεαστεί όλο ο συμβιβασμό αν γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε το All Common Agriculture, μπορεί να υποστηρίξουμε το συμβιβασμό. Διαφορετικά εμείς θα πρέπει να καταψηφίσουμε, αν δεν αφαιρεθεί αναφορά στη Γεωργία, η συγγήτρια. Το, η συμπερίληψη της Γεωργίας, μπορούσα να μιλήσω including agriculture ήταν κάτι που συμπεριλήφθηκε σε πολλές τροπολογίες, συμπερίληψη της γεωργίας, όχι κοινή αγροτικής, η συμπερίληψη της γεωργίας, η λέξη γεωργία. Δεν συμφωνώ με την προφορική τροπολογία. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ο καθένας θα υπομειστεί τις ευθύνες του. Δεν θα ψηφίσουμε κατά τμήματα. Οπότε θα, θα ψηφίσουμε τις προφορικές τροπολογίες και αυτές κυρίως της κυρίας Συντόνια και αντικατάσταση του traditional με τη λέξη fundamental. Παραδοσιακό με θεμελιώδες. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας G λατινικό ως τροποποιήθη. Σας ευχαριστώ. Κατά. Οι φιλελεύθεροι είναι κατά για τους λόγους που μας εξήγησαν. Και η συγγήτρια επίσης. Φιλελεύθερη, πράσινη και γκουε για τους λόγους που εξήγησε ο εκπρόσωπος των τριών ομάδων, ο κύριος Αλβάρο. Ωραία. Συμβιβαστική H, λατινικό. Εδώ ο Γκόραν έχει κάποιο σχόλιο. Εδώ είχα μία προφορική διότι μιλάμε για πολιτική του διαστήματος. Θα πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν ότι δεν στέλνουμε πυράβλους ή κατακτούμε το φεγγάρι, αλλά το ΓΜΕΣ έχει μεγάλη σημασία για τον τομέα του περιβάλλοντος. Μετά τη λέξη technological θα θέλαμε να προσθέσουμε και το environmental. Δηλαδή όχι μόνο τεχνολογική αλλά και ε, πρόοδο υπέρ του περιβάλλοντος. Ναι, πολύ σημαντικό πολιτικά και νομίζω ότι δέχεστε, δέχεται η ΕΛΓΑ την προσθήκη αυτή. Α, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, κανένα λάθος. Η Συντόνια. Η Συντόνια τάσεται υπέρ και η ΕΛΓΑ... Ναι, συμμερίζομαι την άποψη της κυρίας Τρούπελ. Ποιοι είναι υπέρ του ΑΣ όπως έχει τροπήθει από τον Κέραν. Κατά κανείς, όλοι είναι υπέρ του περιβάλλοντος, άρα εγκρίνεται. Αποχή. Ναι. Δεν ρωτήσατε πόσες είναι οι αποχές. Με συγχωρείτε. Καταγράφουμε λοιπόν λοιπόν ότι οι πράσινοι δεν δέχονται το περιβαλλοντικό. Ή κανένας δεν ζητά το λόγο, ποιοι τάσσονται υπέρ, κατά, αποχές, μία αποχή, ο κύριος Πόρτας. Στη συνέχεια έχουμε το, την πρόσυμβασμού G. Ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Όχι, έκανα λάθος. Η συντόνια. Από ό,τι έμαθα, ο κύριος Γκουτμάνης θα ήθελε να αποσύρει την 66. Την 66, άρα αποσύρεται μία από τις προτάσεις του Τζέι και θα σας πω ποια καταπίπτει. 4,5 δισεκατομμύρια από ESF και ERDF για τα έτη 2006-2007. Τα ποσά αυτά δεν ανελήφθησαν από τα κράτη-μέλη και σταματάμε στο Member States, στο J. Εδώ είναι το δεύτερο στοιχείο της ξεχωριστής. Άρα δεν ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα γιατί καταπίπτει δηλαδή αποσύρεται. Άρα δεν υπάρχει ξεχωριστή. Να εξηγούμαστε. Το δεύτερο μέρος καταπίπτει διότι πρόκειται για μια τροπολογία που αποσύρθηκε από τους συντάκτες. Άρα ψηφίζουμε το J που δεν περιλαμβάνει παρά το πρώτο μέρος. Ποιος στάσεται υπέρ. Κατά αποχές. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε στο κάπα. Λατινικό κάπα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελ. Κανείς δεν ζητάει το λόγο υπέρ. Κατά η Χέλγα αντιτίθεται και ο κύριος Πόρτας, αποχές, εγκρίνεται. M, λατινικό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, πόρτας, αποχές, καμία αποχή, εγκρίνεται. N, τροπολογία συμβασμού, N, υπέρ. Σας ευχαριστώ, κατά, κανείς αποχές εγκρίνεται. Ο λατινικό. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ουδής αποχές, ουδής εγκρίνεται. Πι λατινικό υπέρ. Κατά. Δύο αντιτίθενται, αποχές, μία αποχή. Άρα εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις συμβασμού. Σας ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να δούμε τις άλλες τροπολογίες που δεν έχουν απαλληφθεί από τις τροπολογίες συμβασμού. Ένα. Γιούτα Χάουγ που είναι προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οι δύο και οι τρία καταπίπτουν γιατί είχαμε τροπολογία συμβασμού, Τέσσερα, Μπαλτσάνι και Γκέραν. Η συγκήτρια αντιτίθεται. Ποιοι είναι υπέρ. Ωραία ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία και αρχίζει. Για την τέσσερα Πέρας. Δεκαεννέα κατά απορρίπτεται. 5. Βέρτμαν. Η συγγύτητα τίθεται κατά, υπέρ. Ωραία, ηλεκτρονική ψηφοφορία καλύτερα. Ψηφίζουμε την 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται 16 κατά, 13 υπέρ. Άρα ψηφίζουμε την 6. παλσάνι και Φέρμ υπέρ. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπάρχει μία προφορική της εισηγήτριας στο 7. Αντί για internal assessment, own assessment. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Χάουκ 7 εισηγήτρια είναι υπέρ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 Μπιτζότο της κυρίας Μπιτζότο. Αντιτίθεται η συγγήτρια υπέρ. Α, η Μπάρμπαρα είναι υπέρ. Κατά τώρα ψηφίζουμε. Α, τώρα είναι κατά η Μπάρμπαρα. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννέα. Μπαλτζάνι και Φέρμε. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ της εννέα. Η αριστερά. Και πέραν αυτής. Καλά, καλά, καλύτερα ηλεκτρονική. Ο κύριος Άλβαρο ε, δεν δέχεται να συνταχθεί με την αριστερά πέρας. Δεκαπέντε κατά. Δεκατέσσερις υπέρ. Απορρίπτεται. Αρπολογία 10. Τη ελίτ του ΕΛΚ. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Έχουμε την ίδια πλειοψηφία νομίζω λέει ο πρόεδρος. 11. Γένσεν. Αν Γένσεν. Που συμβαδίζει με τη 10. Η σύγητρα είναι υπέρ, υπέρ. Μεγάλη πλειοψηφία κατά. Μικρή μειοψηφία εγκρίνεται. 12, 13, 14, 15, 16 έχουν καταπέσει. Άρα 17. Η συγγήτρια αντιτίθεται υπέρ κατά απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία 18. 18 και 19, αλλά θα πρέπει να ψηφιστούν ξεχωριστά. 18 μπιτζότο, η συγγήτρια είναι κατά, υπέρ, κατά, μειοψηφία κατά, 19, τη σελή του ΕΛΚ, υπέρ, η συγγήτρια είναι υπέρ, κατά, η Χέλγα αποχές εγκρίνεται. 20. που είναι η Ιταλική τροπολογία που στηρίζει η συγγήτρια υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές και η ΧΕΛΜΚΑ. Άρα εγκρίνεται. Άρα 21, 31, 59 καταπίπτουν. Δεν έχουμε ούτε μέχρι την 26. Φτάνουμε στην 27. Άρα έχει, ληφθεί, έχει συμπεριληφθεί. Α, όχι, όχι. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση συμβιβασμού. Στην απολογία συμβασμού. Λοιπόν, 27. Χολμάγερ. Η συγγήτρια τάσεται υπέρ. Υπέρ της 27. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 Χέρτσοκ. Α, καλύπτεται. 29 Βέρτμαν, η συγγήτρια τάσεται υπέρ, υπέρ, ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται 30, Μπιτζότο δεν καλύπτεται, η συγγήτρια είναι υπέρ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 31 των φίλων μας από το ΕΛΚ ε, καλύπτεται. 33. Νέα τροπολογία των Ιταλών. Η συγήτρια τάσεται υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ουδείς αποχές. Βίβα Ιταλία. Εγκρίνεται. 32. Καταπίπτει. 34. Πολυεθνική και πολυκομματική. Η συγκεκριμένη υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά. Οι σοσιαλιστές αλλά είναι απομονωμένοι, άρα εγκρίνεται. 35, 36, 37 καταπίπτουν και η 38 καταπίπτει 39. Η συγκίτρια είναι υπέρ, υπέρ. Της 39. Σας ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40. Η συγκίτρια τάσεται υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 της Γιούτα η οποία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο από το Points Out μέχρι το In This Context. Αντιτίθεται η συγγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Πρέπει να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά πρώτο τμήμα της 41, το οποίο ψηφίζουμε. Πέρας. 15-15 ισοψηφία. Επειδή είναι τροπολογία λοιπόν απορρίπτεται. Στη συνέχεια, στο δεύτερο τμήμα, η συγγήτρια τάσεται υπέρ, υπέρ. Μεγάλη πλειοψηφία, κατά αποχές περνάει. Τρίτο τμήμα, αντιτίθεται η συγγήτρια, τάσεται κατά, υπέρ παρακαλώ. Ωραία. Η ηλεκτρονικά, να δούμε αν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 15-14. Άρα εγκρίνεται το τρίτο μέρος. Ελπίζω το τελικό κείμενο βγάζει νόημα. 42. Χολμάιερ και Βέμπερ. Ε, υπέρ παρακαλώ των Βαβαρών. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η Χέλγα απέχει 45, 45 γιατί καταπίπτουν οι 43 και 44, τρία μέρη, πρώτο τμήμα μέχρι το monitoring, αντιτίθεται η συγγήτρια, ποιοι είναι υπέρ, ηλεκτρονικά καλύτερα ας ψηφίσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα τη 45, πέρας, σας εχουμε έχουμε ισοψηφία 15-15, άρα απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, τάσεται η συγγήτρια υπέρ, όλοι φαίνεται, κατά αποχές. Τρίτο τμήμα, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία και πάλι 15 υπέρ και κατά, άρα απορρίπτεται. Άρα το πρώτο τμήμα απορρίφθηκε τη 45. Άρα ψηφίζουμε τη 46. Μπιτζότο υπέρ, η είναι κατά. Κατά. Όλοι φαίνεται. Γιούτα, Χάουγ, 47. Καταπίπτει, έτσι δεν είναι, γιατί έχουμε απορρίψει το τρίτο τμήμα. Λυπάμαι, Γιούτα. Καταπίπτει. 48. Παλζάνι, Φέρμ, υπέρ, υπέρ και συγγήτρια, υπέρ όλοι, κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια 49, 50 και 51 καταπίπτουν, όχι όμως και οι 52 την οποία ψηφίζουμε. Η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, μεγάλη πλειοψηφία, κατά αποχές εγκρίνεται. 53, 54, 55 καταπίπτουν, όχι όμως και η 56 την οποία ψηφίζουμε. Η συγκίτρια τάσεται κατά, υπέρ παρακαλώ, κατά, Μεγάλη πλειοψηφία, άρα απορρίπτεται. 57. Η συγγήτρια τα στη υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 που συμβαδίζει με την 57. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ελπίζω η ομάδα, η ομάδα της, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα, η 59 έχει ληφθεί υπόψη στην πρόταση συμβάσμου, δεν θα την ψηφίζουμε. 60-61 δεν τις ψηφίζουμε. 62 Γένσεν. Η εισηγήτρια αντιτίθεται. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 12-12, ισοψηφία και πάλι απορρίπτεται. 63, η 63 καλύπτεται. 64 Γένσεν. Εδώ η συγκίτρια τάσσεται υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Όλοι κατά αποχές εγκρίνεται. 65 Γκοντμάνης. Η συγκίτρια αντιτίθεται, ποιοι είναι υπέρ. ομάδα, από ό,τι φαίνεται κατά απορρίπτεται. Η 66 έχει αποσυρθεί. Οι 67 και 68 έχουν συμπεριληφθεί. Φτάνουμε στην 69 της κυρίας Μπιτζότο. Ο Γκέραν κάτι θέλει να πει. Θα θέλαμε να δείτε την 68. Δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτεται από την πρόταση συμβασμού. Νομίζουμε ότι είναι προσθήκη. Τι πιστεύει η συγκήτρια? Νομίζω ότι θίγεται ένα τέτοιο ζήτημα. Ε, αυτό θίγεται όταν ψηφίζουμε την πρόταση συμβιβασμού. Άρα αποφασίζει ο πρόεδρος. Αλλά εγώ ως εισηγήτρια θεωρώ ότι καλύπτεται. Ψηφίστηκε από την ε, τροπολογία συμβιβασμού, άρα καλύπτεται. Τέλος. Ωραία, θεωρούμε ότι έχει καλυφθεί. 69 Μπιτζότο δεν έχει ψηφιστεί. Η συγκήτρια είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Σοσιαλιστική ομάδα. Μειονότητα όμως. Εγκρίνεται. 70 του Λάσλο Σούριαν. Η συγκήτρια είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ποχές εγκρίνεται. 71 καλύπτεται από την ΚΑΠΑ. Η 72 πρέπει να ψηφιστεί η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Δειλά δειλά το ΕΛΚ. Κατά. Αχα. Μάλιστα, διχάζεται λοιπόν το ΕΛΚ. Απορρίπτεται. Η 73 καλύπτεται. Όχι όμως η 74. Σούζια. Η συγκεκριτή είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 75 της κυρίας Μαγκίνες. Προφορική τροπολογία. Ε, δύο φορές θα αντικατασταθεί το 2α από το 2. Τίτλος 2, όχι 2α δεν υπάρχει. Μάλιστα υπέρ της τροπολογίας Μαγκίνες είναι και συμπαθητικό ε, όνομα την ώρα που πρέπει να πιούμε ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνετε εννοώ. Κατά. Αχα, πρέπει να κάνουμε ψηφοφορία ηλεκτρονική. Υπέρ κατά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. υπέρ 16-12 κατά. Μάλιστα, οι 76-77 έχουν καλυφθεί. Οι 78 του Ager είναι κατά η συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ, μόνο η ομάδα του. Καλώς κατά, οι υπόλοιποι. Απορρίπτεται. 79 νέα Ιταλική τροπολογία. Στη συγκήτρια είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές απορρίπτεται. η εισηγήτρια στην 80 τώρα, τα είστε κατά, υπέρ παρακαλώ, κατά, καλώς, ας ε, κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ, στην 80, υπέρ 15-14 κατά, εγκρίνεται, η 81 συμβατή, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 82. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. οντα 83, 84, 85 καταπίπτουν, καλύπτονται δηλαδή. Όχι όμως 86. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Απορρίπτεται η 87 πάλι με τους ίδιους συντάκτες. Η είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά όλοι. Απορρίπτεται. ...89 οι Ιταλοί έχουν σήμερα αποχαλινωθεί τόσες τροπολογίες. Υπέρ, κατά, αποχές, πάλι κερδίζει η Ιταλία. Στην 90 Άλβαρο, σημαντική προσωπικότητα της Επιτροπής μας, ο Χολμάιερ, επίσης σημαντικότητα προσωπικότητα, φυσικά είναι υπέρ η συγγετρία, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, κερδίσατε, μπράβο, 91 Βαλζάνι και Φέρμα, υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 92 με τους ίδιους συντάκτες, ο κύριος Άλβαρο έχει κάτι να μας πει. Ναι, για τους ε, συντάκτες θα θέλω να διατυπώσω μια ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεται αυτή η αναφορά. Στο Εράσμους Μούντους που βρισκεται αυτη η αναφορα στο ερασμος μουντους που αναφερεται για μια υποσημείωση. Θα πρέπει να υπάρχει κάπου στο κείμενο, έτσι δεν είναι. Δεν το βλέπω. Η τρία. Στο αρχικό μου κείμενο, ό, όντως όπως επισημάνατε, υπήρχε το εράσμος Μούντους. Όμως την τροπολογία της κυρίας Βαλτζάνη και του κυρίου Φέρμα ε, απαλήφεται αυτή η αναφορά. Δεν υπάρχει όμως η σαφής επισήμανση μέσα στο κείμενο, μέσα στο έγγραφο, που κανονικά θα έπρεπε να αναφέρεται με τους παχείς, με τους λιπαρούς δηλαδή χαρακτήρες στο αρχικό μου κείμενο. Έτσι είναι κανονικά, έτσι κάνουμε. Λέω, εγώ δεν θέλω να επανέλθω. Σα ευχαριστώ, λέει ο κύριος Άλβαρο, αλλά στην 38 που έχω εγώ, στην έκδοση που μας στείλατε εχθές, δεν βλέπω Εράσμους Μούντου πουθενά. Ναι, σημείο αναφορά όμως είναι η αρχική έκθεση. Εάν δεν υπάρχει τροπολογία για διαγραφή κτλ. παραμένει το αρχικό κείμενο. Oui, autrement euh, ε, για να καταλάβω καλά, εάν ε, κατάλαβα καλά, προτείνεται να διαγράψουμε την αναφορά στο Erasmus Mundus. Ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω να διαγράψω αυτό το σημείο μπορεί να αναφέρεται ε, σιωπηρά αν θέλετε στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων. Πρέπει να μείνει. Και θέλουμε και υποσημείωση για να πούμε ότι αυτό υπάγεται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Μάλιστα, ο κύριος Φέρμ βλέπω ότι συμφωνεί, λέει ο πρόεδρος. Άρα, κατά λάθο διαγράφει εκ παραδρομής δηλαδή το μόνο τους παρελήφθη. Ο James Ellis στη στο λόγο, όχι. Α, όχι, ευχαριστώ πολύ. Συντόνια. Ναι, ε, στο κατάλογο των ψηφοριών υπάρχει μια αναφορά στην συμπερίληψη των ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην 92. Δηλαδή για, τους, ε, για τα άτομα με αναπηρίες λοιπά Έτσι. Η Special Olympics είναι για τα άτομα με πνευματική αναπηρία. Το καταλάβατε όλοι. Εράσμους Μούντους επανέρχεται με τη διόρθωση στην υποσημείωση και τους ε, ειδικού Ολυμπιακούς. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 πόρτας. Η συγκήτρια δεν είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Η συγκήτρια είναι κατά. 94, 95, 96 Καλύπτεται. Πάμε στη 97. Σαλαφράγκα. Μας ξαφνιάσατε. Ε, η συγκήτρια είναι υπέρ όμως. Υπέρ, ευχαριστώ κατά. Εποχές. Ενεκρίθη λοιπόν, όπως είναι οικονομημένος ο συνάδελφος. Στην 98 η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Η είναι υπέρ. Κατά. Οι περισσότεροι άλλοι δυστυχώς απορρίπτεται. Στη συνέχεια, 99, 100, 101, 102 ε, απαλήφονται διότι έχουν καλυφθεί. Στην 103 τώρα η συγκεκριμένη είναι υπέρ. Ευχαριστώ υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται η 104, 105 και 106 καλύπτονται. Μπορούμε να περάσουμε στην 107 του κυρίου Πόρτος Η συγκίτρια τάστε κατά, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Ευχαριστώ αποχές, απορρίπτεται. 108 και πάλι του κυρίου Σαλαφράγκα φαντάζομαι έχει να κάνει με του και πολιτική, υπέρ, συγκεκριμένη, είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 109. Γκουαλτιέρη και λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι κατά. Κατά παρακαλώ, ε, υπέρ παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Γκουαλτιέρη, 109. Αχα, ξαφνικά έγινε μπλε η ψηφοφορία μας, τι διασκεδαστικό αν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε αυτό το... Δεν υπάρχει λόγος για μυστική ψηφοφορία. Εγώ το έκανα το λάθος με τα κουμπάκια. Ναι, βέβαια, η συγγήτρια ένα αμφιβόλο ρίχνει το φταίξιμο στον πρόεδρο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Όχι, δεν γίνεται έτσι ψηφοφορία. Μήπως θα μπορούσε ο τεχνικός να μας μηδενίσει το, το, το σύστημα των ψηφοφοριών. Να ξαναρχίσει η ψηφοφορία. Γκουαλτιέρη, λοιπόν, ξαναρχίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε τη ψηφοφορία και να δούμε μετά ποιο ψηφίζει τι. 18 υπέρ, 11 κατά, Γκουαλτιέρη εγκρίνεται. 110 σαλαφράγκα, η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές. Μπραντνερ 111, είναι κατά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 112 Χαγλουντ. Η είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές. Δεν 113. Χαγνούντ πάλι και Άλβαρο η συγγήτρια όμως είναι κατά πια. Υπέρ παρακαλώ. Μάλιστα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστε τη ψηφοφορία. 16 υπέρ, 17 υπέρ 13 κατά, 114 τώρα της Γιούτα Χαουκ που θέλετε 140 εκατομμύρια να κάνει 135. Προφορική τροπολογία. Α, και Συντόνια, και Συντόνια μάλιστα. Η συντόνια κάνει προφορική τροπολογία. Θα κρατήσει τα 5 εκατομμύρια υπέρ της τροποποιημένης τροπολογίας. Κατά. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Λοιπόν, 115 με την σύμφωνη γνώμη της ηγήτριας υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Εγκρίνεται. 116 της ηγήτριας προσωπική της τροπολογία. Είναι υπέρ βέβαια. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 η είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 πάλι της συγκήτριας. Όλοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική της εισηγήτριας στην έκτη Παύλα, πρόκειται για διαγραφή. Τεχνικού τύπου τροπολογία, όλοι το υποστηρίζουμε έτσι δεν Αποχές εγκρίνεται. Προφορική στο, στην 7η Παύλα με μια προσθήκη λαμβανωμένη υπόψη χρωμοδοτήσεως της Επιτροπής Αναπτύξεως. Η συγκεκριμένη είναι υπέροχη, από φαίνεται. Εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε το σύνολο της εκθέσεως, όπως τροποποιήθηκε παρακαλώ. Υπέρ, ευχαριστώ, κατά, αποχές, κανένας. Τέσσερις αποχές. Τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση, συγχαρητήρια στη Σιδόνια και ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους. και ζητούμε συγγνώμη για τα προβλήματα με το κείμενο, με τη μετάφραση και χρειάστηκε να είμαστε ευέλικτοι. Τώρα έχουμε την τελευταία ψηφοφόρια. Αφορά την έκθεση της Γιούτα πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τροποποιώντα τον κανονισμό του Συμβουλίου για τι δομέ για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματο και Προγράμματο Ραδιοπλοήγηση. Για το Γαλιλαίο, με άλλα λόγια. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορία όλοι και το ΕΛΚ. μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδικά. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να ψηφίσουμε ομαδικά κάποιες τροπολογίες. Ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα την πρόταση ψηφίσματος, νομοθετικού ψηφίσματος, υπέρ, κατά, αποχές, ομοφωνία. Εν συνεχεία, όσον αφορά την νομοθετική πράξη αυτή καθεαυτή, τέσσερις τροπολογίες λοιπόν της Ιούτα μαζί υπέρ, κατά ουδείς αποχές, καμία αποχή, θρίαμβος, πρόκειται περί θριάμβου. Ε, συγχαίρουμε λοιπόν τη Γιούτα. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. είχαμε βάλει και ενδεχόμενες μεταφορές στο σημείο 14 και 15, όμως, ας το επιβεβαιώσουν αυτό οι συγκητές, δεν υπάρχει αίτημα μεταφοράς τελικά. Άρα δεν έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Schengen, το σύστημα δεύτερης γένειας. Έχουμε έναν εισηγητή, τον κύριο Αλβάρο, και έχουμε τα σημεία 7 και 8 σχετικά με το θέμα αυτό. Θέλουμε να τροποποιήσουμε έναν κανονισμό και μία απόφαση του Συμβουλίου. Αλεξάνδρ, παρουσιάστε εντάχει το θέμα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, γιατί τα σημεία 7 και 8 είναι ταυτόσιμα προς το κείμενο. Ε, το έχει η Επιτροπή των Ιστορικών αυτή τη στιγμή προς εξέταση το ζήτημα. Εμείς και η συνάδελφος Χολμάιερ βέβαια και εγώ έχουμε και ο κύριος Διακόπτει ο μιλητής. Τόσο σύντομα, Πρόεδρε, τόσο σύντομα. Λίγο χρόνο δώστε μου τουλάχιστον. Λογοκρισία, έτσι. Λοιπόν, ας είμαι σύντομος. Δεν έχω και πολλά να πω για το θέμα. Είναι ένα θέμα λοιπόν της Επιτροπής των Ιστορικών, εισηγητής είναι ο κύριος Κοέλιο. Έχουμε ε, συνομιλήσει μαζί του, βλέπουμε ικανοποιητικέ ε, προτάσεις, έξι μόνο είναι δικές μας τροπολογίες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και προτείνουμε για το προπολογισμό του 2011 τα ποσά για το σύστημα ενημέρωσης Σέγγεν στη δεύτερη, της δεύτερης γενεάς να πάνε στο αποθεματικό και να αποδεσμευθούν όταν μπορεί να εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο συγκεκριμένα τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και μπρος. 70 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε περίπτωση. και θα πρέπει να διαρευνήσουμε ε, αν θα λειτουργήσει τον, η νέα τεχνολογία με το Frontex κτλ. Αυτά λοιπόν, όπως είπα, θεματικό για τα ποσά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τις ε, προόδους και για τα ε, εμπόδια, τις δυσκολίες που διαπιστώνονται μπορούμε πιστεύω να βελτιώσουμε ουσιαστικά την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο ακόμη από ό,τι στα προηγούμενα χρόνια και ταυτόχρονα σημειώνουμε ότι επιδιώκουμε μια αποτελεσματική εναλλακτική για το δεύτερη γενεά του SIS γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής λειτουργήσει ικανοποιητικά. Και σημειώνουμε επίσης ότι δεν θέλουμε επιπλέον επιβάρυνση, οικονομική επιβάρυνση με το νέο σύστημα. Το καταγράφουμε με τις τροπολογίες μας. Αυτά νομίζω μπορούμε να είμαστε σύντομοι. 12 Μαρτίου είναι η προθεσμία για την καταθέση των τροπολογιών. 16-17 νομίζω μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. 7-8 Απριλίου στην Επιτροπή των Ιστορικών ε, θα γίνει η ψηφοφορία. Πάντως ήθελα να επισημάνω ότι τις τροπολογίες έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει με τον συγκεκριτή τον κύριο Κοέλιο. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ασφαλώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα. Έχουν να κάνουν και με τον έλεγχο και την ασφάλεια των εισόδων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Κύριε Χολμάιερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ τάσσομαι επικριτικά εναντί αυτού του θέματος. Δεν μπορώ λοιπόν να δηλώσω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τις μέχρι τώρα εξελίξεις στο σύστημα του SIS. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε επεξεργαστεί επί χρόνια. Πολλά χρήματα έχουν διατεθεί. Κάποια ζητήματα έχουν ενδεχομένως προκαλέσει ερωτηματικά που πάνε πια χρήματα, πια ποσά. Θα πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Χρειάζεται ένα σύστημα κατεπηγόντως να τεθεί σε ισχύ γιατί δεν υπάρχει ούτε η διαφάνεια, ούτε η επικοινωνία που θα θέλαμε. Και ελπίζω ότι μετροπολογίε Γιατί πιστεύω ότι οι αλλαγέ αυτέ θα γίνουν σχετικά σύντομα πάνω απ' όλα, γιατί θα πρέπει να αποφασίσει τον Απρίλιο το Συμβούλιο. Και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με τις υφιστάμενες συνθήκες. Άρα είναι η πίεση του χρόνου αρκετά σημαντική. Η Επιτροπή κάνει κάποιες δηλώσεις ε, σαν να θεωρεί ότι τα πάντα ήταν απόλυτος επιτυχημένα. Φαίνεται ότι κάποια κράτη-μέλη όμως όντως δεν βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και βλέπουν ότι τα χρήματα δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως τα έπρεπε. Ίσως να βρούμε λύσεις διαφορετικές από τις 26 ώρες, παραδείγματι. Υπάρχουν στη χώρα μου, εφερειπίν, ε, ε διαπιστώσω ότι οριστικά δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα, έχει καταρρεύσει συνολικά και έτσι χρειάζεται αλλαγή αντικατάσταση. Ίσως λοιπόν ε, θα χρειαστεί, Πρόεδρε, να συζητήσουμε και να έρθουμε σε αντιπαράθεση με το, ως προς το θέμα αυτό και με την Επιτροπή των Εσωτερικών. Δεν είναι καλό, ύστερα από 8 χρόνια δοκιμών και επιχειρήσεων ε, με ένα ηλεκτρονικό σύστημα, να μην είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι σε θέση να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είμαστε και σοβαροί έναντι των άλλων εταίρων με τους οποίους καλούμεθα να συνεργαστούμε. Euh, euh, Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω Ε, το σύστημα Schengen, ξέρετε, ξεκίνησε πριν να κοινοτικοποιηθεί. Μάλλον ξεκίνησε το σύστημα πληροφοριών πριν να κοινοτικοποιηθεί το, το Schengen. Λοιπόν, τότε ήμασταν 7-8 χώρε Schengen ε, από, τις 12, από τα 12 κράτη-μέλη και αποφασίσαμε τότε να, να ετοιμάσουμε την πρώτη εκδοχή του συστήματος του ε, πληροφοριακού της, του Schengen. Και τότε δεν λειτουργούσε και ήδη είχαμε επικρίνει πολύ το σύστημα που έχει επιλεγεί. Δεν ήταν τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ήταν αρμόδια ακόμα, υπήρχε μια εκτελεστική γραμματεία και ήταν ένα σύστημα καταστροφικό εντελώς. Και αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική κατάσταση διότι αντιμετωπίζουμε τεχνικό πρόβλημα που είναι λίγο δύσκολο αλλά τώρα έχουμε περίπου 10 χρόνια εμπειρίας και δεν βρήκαμε πάντα ικανοποιητικές λύσεις ακόμα και εντός του κοινοτικού πλαισίου. Όμως είναι θεμελιώδες εργαλείο για την προστασία των εξωτερικών μας ε, συνόρων. Και γνωρίζουμε ότι το μοντέλο αυτό το ευρωπαϊκό υποθέτει ότι μπορούμε να συνδυάσουμε την προστασία των πολιτών εναντί τρομοκρατίας, μαφίας κλπ και ταυτόχρονα την προστασία των ατομικών ελευθεριών. Αν δεν έχουμε τα τεχνικά εργαλεία για να το πετύχουμε αυτό, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ε, απογοητευτικό για την Ένωση. Δεν ξέρω αν θέλετε, θέλεις Αλεξάνδρ να προβεί σε κάποια σχόλια. Σας ευχαριστώ όπως είπε και εισηγητής όσον αφορά τα δύο κείμενα που είναι σχέδιο κανονισμού ε, από τη μια και σχέδιο αποφάσεως από την άλλη θα γίνει ψηφοφορία στις 16 και 17 Μαρτίου η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή 7 και 8 Απριλίου και στη Σύνοδο του Απριλίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Είχαμε άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη η συνέχιση της ζητήσεως επί της εκθέσεως του κ. Γκολτμάνης, αλλά ο κ. Γκολτμάνης ε, απουσιάζει, ζητά συγγνώμη γι' αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπων με τον οποίο είχε εμπλακεί στο θέμα προσωπικά και στην έκθεση, θεωρώ ότι δεν θα ήταν ευκταίον να διεξαχθεί συζήτηση σαν αυτού. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι που μείνατε μέχρι το τέλος, η αριστερά εξαφανίστηκε από την Επιτροπή Προπολογισμών. Γκόραν την οικία. Όχι, όχι, Γκόραν, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Γκόραν. Όχι, όχι, όχι, όχι, σε πείραζα, πείραζα, πείραζα. Από τη συνάδελφη, σε ευχαριστώ πολύ. Εξατλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Στους συντονιστές προτείνω να παραμείνουν εντός εθούσης να ακολουθεί συνεδρία συντονιστών αμέσως και να εκμεταλλευτούμε την παρουσία των διερμηνέων, τους οποίους ευχαριστώ, ούτως ώστε να διεξαχθεί συνεδρίαση των συντονιστών. Λήξη της συνεδρίασης.